Καλησπέρα σας. Μόλις ε, πέρασε και το ακαδημαϊκό τέταρτο, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτή την απογευματινή δευτεριάτικη συνεδρίασή μας και να δούμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω το σημείο 7 με θέμα την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης με συντάκτη γνωμοδότηση τον κύριο Γιάκοφτσιτς αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Όχι, οπότε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες με εξαίρεση τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και εγώ, εδελικά και ελτικά. Και περνάμε στο πρώτο κύριο θέμα της ημερήσια διάταξης που θα μας απασχολεί στο μεγαλύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας και που αφορά ένα εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τη σχέση μεταξύ των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Ο κύριος Δεκάστρο είναι ο εισηγητής μας για το θέμα αυτό. Πριν όμως περάσουμε στην εξέταση της έκθεσης του κυρίου Δεκάστρο, θα ακούσουμε ένα καλεσμένο μας που είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρόκειται για τον κύριο Τομάσο Βαλέτη, καθηγητή, που θα μας μιλήσει για τον πιθανό αντίκτυπο της έγκρισης νομοθεσίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ο τίτλος της παρουσίας του καθηγητού Βαλέτη αφορά τη ρύθμιση των τα θέματα των εμπορικών πρακτικών και τον οικονομικό αντίκτυπο στους γεωργούς, μεταποιητές, ε, εμπόρους ελληνικής και καταναλωτές. Μάλιστα, η πρόταση για την παρουσίαση αυτή έγινε από την ίδια την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και το Γενικό Διευθυντή Μαγκέλα. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Βαλέτη. Καλώς ορίζω και τα μέλη της Επιτροπής, φυσικά και τα, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας δίνω το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα αξιότιμα μέλη. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα και που μου δίνεται η ευκαιρία να σας εξηγήσω την τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής. Να σας συστηθώ πρώτα απ' όλα. Λέγομαι το Μαζό Βαλέτη. Είμαι αυτή τη στιγμή επικεφαλής ε, οικονομολόγος στην Digicom. Η κανονική μου δουλειά, ωστόσο, είναι ακαδημαϊκός. Είμαι καθηγητής οικονομικών στο ε, Πανεπιστήμιο της Ρώμης Βεργάτα στην Ιταλία και στο London School of Economics. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τις βασικές ιδέες, τις οποίες γνωρίζετε η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται σε πολύ ε, απλούς πυλώνες. Ο κοινό για όλους μας ε, σκοπός εδώ στην αίθουσα είναι να προστατεύσουμε τους μικρούς αγρότες από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω η πρόταση εστιάζεται απευθείας ε, στα προβλήματα που υπάρχουν. Η νομική βάση είναι σαφής. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μικρούς αγρότες ε, και να τους προσφυλάξουμε από τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές. Η πρόταση έχει δομηθεί έτσι ώστε κάθε φορά που εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα να προτείνεται μια λύση. Όταν όμως τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα, ούτε υπερβολικά σημαντικά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει να υπερβεί τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνει ένα βήμα πίσω, αφήνοντας τα κράτη-μέλη να προτείνουν λύσεις καταλληλότερες για τις ε, τοπικές συνθήκες. Βασικό στόχος της πρότασης είναι να εξευρεθούν κάποιες σαφείς κατευθυντήρες γραμμές. Γι' αυτό επικεντρώνεται κατακόρυφα πρώτα απ' όλα στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, business to business, μεταξύ των γεωργών, των πολιτών και των μεγάλων σούπερ μάρκετ, των αγοραστών. Εκεί εστιάζεται, εστιάζεται και σε τομείς όπου υπάρχει οικονομική ανισορροπία, όπου υπάρχει κάποιο εμπορικό πλεονέκτημα της μίας πλευράς, δηλαδή στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων και η πρακτική πρόταση διάκρισης των μικρών και των μεγάλων βασίζεται σε εκατόφλια τα οποία βασίζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι αδιαφεσβήτητες και αποδεκτές σε ολόκληρη την Ένωση. Επίσης προτείνει να υπάρχει μια μαύρη λίστα πρακτικών που σίγουρα είναι επιβλαβείς. Αυτό αφορά ε, μια μαύρη λίστα, οι οποίες θα απαγορευτούν. Και μετά υπάρχει μια σειρά πρακτικών σε μια γκρίζα λίστα, ανάλογα με τις συνθήκες. Δηλαδή, αυτές ε, οι πρακτικές μπορεί να είναι μαύρες ή λευκές και τι είναι αυτό που καθιστά μια πρακτική κατάλληλη να μπει στη μαύρη λίστα, κατά πόσο έχει γίνει κατανοητή ε, και αποδεκτή από τις δύο πλευρές. Αν αυτό δεν συμβαίνει, μπαίνει στη μαύρη λίστα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα προμήθεια τροφίμων, η οποία είναι περίπλοκη. Γεωργοί, μεταποιητές, ε, λιανοπολιτές, καταναλωτές ε, και εστιαζόμαστε εδώ στον πιο αδύναμο κρίκο, στους μικρούς αγρότες οι μικροί αγρότες, ειδικότερα όταν επηρεάζονται άμεσα από αθέμητε εμπορικές πρακτικές, όταν για παράδειγμα ένας μεγάλος αγοραστής θέλει να επιβάλλει ε, εξοντοτικές ε, συνθήκες ε, σε ένα μικρό γεωργό, υπό πολλέ προϋποθέσεις είναι δύσκολο να τι εντοπίσει κανένα. αλλά υπάρχει και περίπτωση το θύμα μια τέτοια πρακτική να μην είναι ο γεωργό άμεσα, αλλά έμεσα. Ε, να είναι, υπάρχει δηλαδή κάποιο άλλο ε, θύμα το οποίο μεταβιβάζει ουσιαστικά το, ε, τη ζημία στον γεωργό. Η πρότασή μας λοιπόν θα πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι πολύ ρεαλιστική. Διότι θέλουμε να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι εφικτή. Αυτό είναι το δυνατό σημείο αυτής της πρότασης. Ποιον θα προστατεύσουμε? Τους μικρούς αγρότες. η νομική βάση διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης βάσει των προτύπων της ΚΑΠ. Αυτή είναι η νομική βάση. Αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε. Έγινε μια πρόταση επέκτασης ε, του πεδίου εφαρμογή ε, των, των πρακτικών, ε, αλλά σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σα σε πιθανέ ανεπιθύμητε ε, συνέπειες ότι η απαγόρευση ορισμένων πρακτικών μπορεί να μην έχει κανένα όφελος ε, στο ε, κοινό στόχο μας που είναι μικρή γεωργή. Οπότε εστιαζόμαστε κυρίως στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κυρίως μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Εκεί επικεντρώνεται η πρότασή μας γιατί να μην το επεκτείνουμε στι σχέσει μεγάλων επιχειρήσεων, μεγάλων αγροτών και μεγάλων αγοραστών, μεγάλων πολιτών και μεγάλων αγοραστών, μεγάλων σούπερ μάρκετ. Να σα δώσω ένα παράδειγμα για εδώ. Εδώ. Φανταστείτε μια μεγάλη επιχείρηση όπως η Unilever, μια πολυεθνική που διαπραγματεύεται κάποιες προϋποθέσεις με το Σόι, το Ντελέζ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ για ας πούμε παγωταχωνάκια εάν παρέμβουμε ε, στο πλαίσιο μιας αθέμητης εμπορικής πρακτικής ε, ενώ μιλάμε για δύο μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλα περιθώρια κέρδους με διαφορετική δραγματευτική ισχύ ε, αν δεν αφήσουμε δηλαδή την αγορά να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη λύση αν εμείς παρέμβουμε δηλαδή στο πλαίσιο των αθέμητων εμπορικών πρακτικών θα επιτύχουμε το στόχο να προσφέρουμε δηλαδή ένα όφελος για έναν αγρότη στο Βέλγιο που παράγει μεγάλα ο γαλακτοπαραγωγός ο Βέλγος δηλαδή θα κερδίσει κάτι αν ας πούμε αυξηθεί ε, προς όφελος της Unilever η τιμή του παγωτού χωνάκι. Όχι, δεν θα περάσει κάποιο όφελος στον αγρότη. Από την άλλη, αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια σε περίπτωση που κάνουμε κάτι τέτοιο και ανεβάσουμε την τιμή του παγωτού χωνάκι είναι ότι εμείς ως καταναλωτές, ως πολίτες θα καταλήξουμε να πληρώνουμε περισσότερο για αυτό το παγωτό. Αν φυσικά τον τελέζει το Καρφούρ προσπαθεί να διαπραγματευτεί άμεσα με τον Γιώργο, με τον Βέλγο Γιώργο, εκεί καλύπτεται από την πρόταση που συζητάμε εδώ. Παρομοίως, εάν η Unilever λόγω αυτής της UTP σε συναλλαγές επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων προσπαθήσει να διαβιβάσει τη ζημία της στο Γιώργο και αυτό θα καλύπτεται από την πρόταση αυτή, από την οδηγία αυτή. Ε, εστιαζόμαστε λοιπόν, όπω είπα, εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα και δεν κάνουμε κάτι εκεί που θεωρούμε ότι είναι αρκετά μεγάλη παίκτη, ώστε να μην, ε, είναι... να μην προκαλείται τεράστια ζημιά. Ορισμένοι έχουν επίση ε, προτείνει να καθορίσουμε την, σε επεμβάσει μα βάση τη έννοια τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, όπω ξέρετε, είναι μια καταπληκτική έννοια. Η Κομισιόν το αναφέρει συνέχεια και η Επιτροπό μου το αναφέρει συνέχεια στι ομιλίε τη. Η δικαιοσύνη επίσης σχετίζεται και με τον ανταγωνισμό σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερικανική Αρχή Ανταϊτράστα την ονομάζει την τρίτο ε, ονομάζεται ως ε, έχει μια επιτροπή συγγνώμη, ε, του δίκαιου εμπορίου. Υπάρχει αυτή η έννοια του δίκαιου εμπορίου που συνάδει με τον ανταγωνισμό. Στην πρακτική όμως δεν είναι εύκολο να καθοριστεί η έννοια αυτή τη δικαιοσύνη. Του δικαιομπόριο, υπάρχουν διάφορες απόψεις και η υλοποίηση δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί κανείς να κάνει μια ανάλυση κατά περίπτωση και να ορίζει το δικαιομπόριο ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά αυτό είναι χρονοβόρο. Επίση, μπορεί να έχει ανεπιθύμητε συνέπειε για τον παραγωγό. Αν αρχίσουμε να συζητάμε τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο μεταξύ των μερών και αν βάλουμε και τα μέρη να το συζητάνε, το πιθανότερο είναι ότι οι δυνατότεροι, οι μεγάλοι αγοραστέ, θα έχουν περισσότερου οικονομικού πόρου για να επηρεάσουν τη διαδικασία και πάλι δεν μπορούμε εδώ να προστατεύσουμε του μικρού αγρότε. Οπότε το να μπούμε σε μια συζήτηση του τι είναι δίκαιο, ενώ είναι ενδιαφέρον θεωρητικά, μπορεί να οδηγηθούμε σε προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή. Παραμένουμε λοιπόν πολύ ρεαλιστές και γι' αυτό το λόγο επικεντρωνόμαστε σε ένα σύνολο καλά καθορισμένων επιβλαβών πρακτικών, αναποτελεσματικών, αλλά χωρίς να θέλουμε να υπερβάλλουμε. Μπορώ να σας δώσω δύο παραδείγματα εδώ που είναι ενδιαφέροντα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος ε, γεωργός είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, έχει επινοήσει ένα νέο προϊόν το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα στην αγορά κάποιο υβριδικό προϊόν μεταξύ ροδάκινων και δαμάσκινων ε, και ροδάκινων και βερίκοκων, συγγνώμη Μπορεί να θέλει λοιπόν ο Γιώργος αυτός να δώσει κάποια κίνητρα στους ε, πολιτές για να βάλουν αυτά τα προϊόντα στα ράφια τους. Υπάρχει κάποιο κίνδυνος εκεί. Μπορεί να θέλει δηλαδή να συμμετέχει και στην προώθηση του προϊόντος αυτού, το οποίο πιστεύω ότι είναι καλό και θα πρέπει να μπει στην αγορά, αλλά θα πρέπει να δοκιμαστεί. Αν εμεί πάμε και πούμε ότι τέτοιε εκστρατείε πρόθεση, ε, ε, σε αυτέ τι εκστρατείε πρόθεση δεν πρέπει να συμμετέχουν οι γεωργοί, η κακή πλευρά το πρόβλημα θα είναι ότι μετά ο αγοραστή, ο λιανοπολιτή μπορεί να μην θελήσει να δεχτεί αυτά τα προϊόντα καθόλου. Υπάρχει υπερβολικό κίνδυνο. Οπότε εκεί επιτυγχάνουμε το αντίθετο, ότι ο μικρό γεωργό που καινοτόμησε και ε, το ρηψοκινδύνευσε δεν θα μπορέσει να πουλήσει τα προϊόντα του. Τα προϊόντα αυτά δεν θα φτάσουν στους καταναλωτές. Όπως είπα νωρίτερα, υπάρχει μια μαύρη λίστα περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της ε, πρότασης οδηγίας. Και υπάρχει και μια γκρίζα λίστα. Η γκρίζα λίστα, κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να την αφήνουμε στη διακριτική ευχαίρεια των ε, φορέων. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο κατόφλιο για μια πρακτική που θα λέει ότι μετά από αυτό το κατόφλιο γίνεται δεκτή ή όχι ε, οικονομική ορολογία λέμε εξάντε και exposed. Εάν λοιπόν η πρακτική είναι δεκτή μεταξύ δύο συμβαλόμενων μερών του Γεωργού και του αγοραστή, τότε είναι εντάξει. Αν είναι exposed, εκτεθειμένη, δηλαδή αν εκπλήσει ξαφνικά ή στραγγαλίζει το Γεωργό, αν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες ε, ε κινδύνου που θα διαβιβαστούν στο Γεωργό, αυτές τις πρακτικές θέλουμε να αποφύγουμε και να απαγορεύσουμε ώστε να αποφύγουμε ανεπιθύμητες συνέπειες. Αυτό θα πρέπει να ρυθμίζει λοιπόν η οδηγία. Δεν σχεδιάζεται στο πλαίσιο τη οδηγίας να ρυθμίζονται και άλλες πτυχές. Τιμές, για παράδειγμα, μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών. Δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε τιμές. Δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σχετικό κόστο, Σε μεγάλο βαθμό ε, ζούμε σε μια οικονομία αγοράς, οπότε η ε, ε, παροχή και η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν επενδύσεις και τις τιμές. Εάν εμεί παρέμβουμε σε αυτόν τον μηχανισμό, μπορεί να οδηγήσουμε σε κατάρρευση του οικονομικού συστήματος. Παρορισμένες προτάσεις που έχουν γίνει δεν ε, προτείνουμε να ρυθμίσουμε τιμές λιανικής. Δεν είναι αντικείμενο αυτό αυτής της οδηγίας. Αναφέρεται και στην εκτίμηση αντικτύπου. Δεδομένων αυτών, στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης έχουν γίνει καλόπιστες προσπάθειες ρύθμισης των ε, λιανικών τιμών και αυτές οδήγησαν σε ανεπιθύμητες συνέπειες που εμείς δεν θέλουμε σήμερα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία είχαμε τον ε, νόμο Γκαλάν περίπου πριν από 8 χρόνια ναι με τον οποίο καλόπιστα έγινε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τα μικρομάγαζα από το μεγάλο ανταγωνισμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η πρόθεση δηλαδή ήταν καλή. Αλλά αυτό που έγινε τελικά ήταν ότι δεν άφηναν τις τιμές να πάνε κάτω από το κόστος με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι τιμές λιανικές ανέβηκαν υπερβολικά. Ε, τα περιθώρια κέρδου λοιπόν των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν υπερβολικά και δεν υπήρχε κανένα όφελο για τα μικρομάγαζα. Αυτό έγινε κατανοητό και μετά ε, καταργήθηκε όμω αυτό και συνέχισε να λειτουργεί η οικονομία ω οικονομία τη αγορά. Συνοπτικά λοιπόν, οι κύριοι πυλώνε αυτή τη πρόταση είναι οι εξή. Ε, επιχείρηση προ επιχείρηση, business to business. Σχέσει μεταξύ αγοραστών και γεωργών δεν ρυθμίζουμε τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η πρόταση επίση ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ μικρών και μεγάλων. Εκεί παρατηρούνται οι οικονομικέ ανισορροπίε. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε να καθορίζεται η σχέση ε, βάσει μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα υπάρχει και κάποιο κατόφλιο αναγνωρισμένο σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει το κατόφλιο αυτό να θεωρείται και δίκαιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το, τις πρακτικές, ε, το αντικείμενο, Κάποιες πρακτικές ε, εξετάστηκαν ε, στην εκτίμηση αντικτύπου και αποδείχθηκαν κακές, ε, μπήκαν στη μαύρη λίστα και άλλες πρακτικές μπορεί να είναι ή όχι επιβλαβείς, ανάλογα με το κατά πόσο έχουν γίνει κατανοητοί και είναι σαφείς οι συμβατικοί όροι μεταξύ των μικρών γεωργών και των αγοραστών. Αυτός είναι ο κοινό παρανομαστής μεταξύ όλων των κρατών μελών. Γνωρίζουμε ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να θελήσει να ρυθμίσει λίγο διαφορετικά την κατάσταση λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας δεν απαγορεύει κάποιο σε οποιαδήποτε χώρα να είναι πιο αυστηρή αν, θεω, το θεωρήσει απαραίτητο. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι επαρκής ε, και λογική. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για την παρουσίαση αυτή. Ε, πρώτα θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Δεκάστρο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του και μετά θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές με περιορισμένο χρόνο. Πρώτα ο κύριος Δεκάστρο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο το Μάζο Βελέτη για το πώ συνέβαλε στη συζήτησή μα σήμερα. Είναι καθοριστική εβδομάδα αυτή γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μα. Ταυτόχρονα με τη συνεδρίασή μας τώρα οι συνάδελφοι της, Κομισιό, της Επιτροπής ΙΜΚΟ ψηφίζουν αυτή τη στιγμή τη δική τους γνωμοδότηση οπότε θα πρέπει να δούμε, αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία αυτή. Θα πρέπει να πω στον κύριο Βαλέτη ότι το έγγραφο του που σχετίζεται με την εκτίμηση αντικτύπου για την πρόταση χρησιμεύσε ω οδηγό για να συντάξουμε το σχέδιο έκθεση το οποίο συντάξαμε εμεί. Καθώς επίσης και για πολλέ από τι τροπολογίε που παρουσίασαν οι συναδέλφοι εδώ στην Επιτροπή. Και θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι η δική μας Επιτροπή δεν θέλει σε καμία περίπτωση να περιορίσει τη συμβατική ισχύ των διαφόρων φορέων εντός της αλυσίδα. Εφόσον όμως η ε, ε, δύναμη που έχουν ασκείται με τίμιο και δίκαιο τρόπο. Και εκεί θα πρέπει να παρεμβαίνουμε νομοθετικά. Είμαι βέβαιο ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι μια άριστη αφετηρία. Είναι αναγκαίο να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ε, έχουμε 20 ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όλη η εκτίμηση αντικτύπου έχει τεκμηριωθεί πλήρως. Δεν έχουμε, έχουμε συζητήσει πλέον εκτενώς στην Επιτροπή μας, έχουν γίνει διάφορες συνεδριάσεις με τους κοιόδης, έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Δεν θα μπω στην ουσία, θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο. Ότι η, η μελέτη του δικού μας κοινού κέντρου ερευνών και που προσαρτάται στο σημείο C της εκτίμησης αντικτύπου ε, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο οι κριτικές που συχνά λαμβάνουμε σε σχέση με μια πιθανή αύξηση των τιμών λιανικής ε, ανάλογα φυσικά με τις εθνικές νομοθεσίες φυσικά που προσπαθούν να αποτρέπουν τις αθέμητες ε, πρακτικές. Η φόβη αυτή λοιπόν είναι αβάσιμη τι λέει εδώ αυτός ο πίνακας που είναι πολύ ενδιαφέρον όπως προσαρτάται στη μελέτη αντικτή που μας παρουσίασε ο καθηγητής. Λέει ότι εκεί όπου υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες που περιορίζουν τη συμβατική ισχύ, ισχύ το, αποφεύγοντας τις πρακτικές, εκεί λοιπόν δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση των τιμών λιανικής. Αντιθέτως, στις χώρες όπου υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, οι τιμές λιανικής φαίνεται να αυξάνονται λιγότερο από ότι αυξάνονται στις χώρες όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Οπότε θα ήθελα να μα κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, αν έχετε τη δυνατότητα κύριε Βαλέτη, αν και πώς η οδηγία αυτή που ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε και που ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε εντό τη Αυστριακή Προεδρία θα μπορέσει να βοηθήσει όλου του φορεί τη αλυσίδα για την αποφυγή των αθέμητων πρακτικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα. Να δώσουμε στο λόγο στην κυρία Μάκεντάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίασή της και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Ντικάστρο, για όλη του την ε, μέχρι τώρα εργασία, για την προετοιμασία της έκθεσης αυτή για τις αθέμητες πρακτικές. Πρέπει να υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ε, τροπολογιών. Έχει γίνει πολλή δουλειά και πραγματικά φτάσαμε σε συμβιβασμούς που δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο πόσο καλή ήταν η διαπραγμάτευση. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ξέρω ότι θα ψηφιστεί πολύ σύντομα. Όσον αφορά τώρα τις αθέμητες πρακτικές, εξορισμού πρόκειται για κάτι το αθέμητο. Αυτό το διαβάζουμε ακόμα και στον τίτλο. Άρα, Γι' αυτό και βλέπω εδώ ότι ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε σε κάποιες από τις αθέμητες πρακτικές και όχι σε κάποιες άλλες. Είτε είναι μεγάλος, είτε μικρός αν θέλετε ο προμηθευτής, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε αθέμητες πρακτικές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να επεκτείνουμε λίγο το πεδίο και τον ορισμό, παραδείγματο χάρη να ενσωματώσουμε και άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη τα λουλούδια, εξίσου ε, αναλώσιμα και αλλοιώσιμα είναι τα λουλούδια, όπως ακριβώς και τα φρούτα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να πλησιάσουμε στους ορισμούς μας, στους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και είμαι εξαιρετικά περήφανη γιατί στη χώρα μου έχουμε έναν κώδικα που αφορά όλα αυτά τα προϊόντα γεωργικά και τρόφιμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Κάθε φορά που συζητούμε με ενώσεις ε, παραγωγών, ε, με υπεύθυνους για το λιανικό εμπόριο, Ξέρω ότι αυτός ο κώδικας πραγματικά άλλαξε σημαντικά την κατάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν να επεκτείνουμε αυτή την προστασία και σε άλλους γεωργούς, σε όλους τους γεωργούς δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη και με μεγάλη χαρά θα δούμε αυτές τις πρακτικές να επεκτείνονται. Βέβαια δεν είναι τέλεια η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω ότι είναι μια βάση αρκετά καλή, στην οποία μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε και να στηριχτούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κατάινε. Kiitoksia Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση που μας έκανε. Και εγώ ως σκέφτης ανησυχώ για την πρόταση επέκτασης οδηγίας. Δεν έχουμε μελέτη αντικτύπου για την επέκταση οδηγίας προκειμένου να καλυφθούν και οι υπηρεσίες των γεωργικών προϊόντων. Έχει γίνει κάποιο είδους μελέτη ενδεικτύπου για το θέμα αυτό. Επίσης, έγινε η πρόταση επέκταση οδηγία στο πεδίο εφαρμογή ώστε να καλύπτονται όλοι οι προμηθευτέ. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα. σε περίπτωση που μια, ένας παραγός που είναι πολυεθνική, που πουλά σε, άλλο, σε άλλη πολυεθνική, ε, τι θα γίνει. Το άρθρο 43 ε, σκοπό έχει την εξασφάλιση αξιοπρεπούς γεωργικού οδημάτο για το γεωργό, όχι για την πολυεθνική. Μήπως λοιπόν η επέκταση του πεδίου εφαρμογής ε, θέσει σε κίνδυνο το σύνολο της οδηγίας και διακυβεύσει και την θέση ισχύ της. Ο κύριος Κάρθη που είναι απουσιάζει. Κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για την πρόταση της. Πρόκειται για ένα τομέα που είναι πολύ σημαντικό να τον ρυθμίσουμε. Πρόκειται για θέμητες πρακτικές που οδηγούν σε πολύ σημαντικές τρευλώσεις της αγοράς. Πλήττονται παραγωγή και χαίρομαι ιδιαίτερα εδώ γιατί επεκτείναμε σε ένα σημαντικό βαθμό το εύρος ε, της εφαρμογής, όπως παραδείγματος χάρη συμπεριλαμβάνοντας και τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης γιατί συμπεριλάβαμε και τους συνεταιρισμού. Υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί, πολλές οργανώσεις παραγωγών μέσω των οποίων μπορούν να δράσουν και να ενεργοποιηθούν οι παραγωγοί με διάφορες μορφές εξάλλου περιορισμένης ευθύνη, συνεταιρισμοί, οργανώσεις ε, ε, παραγωγών και ενώσεις ε, συνεταιρισμών. Πιστεύω επίσης ότι κάθε δύο-τρία χρόνια, μπορούμε να δούμε ακριβώς ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να γίνεται ένα είδος παρακολούθησης, monitoring, να δούμε παραδείγματο χάρη αν πρέπει να μπουν καινούριε εταιρείε στη μαύρη λίστα ή να βγουν κάποιες, αν δηλαδή υπάρχουν ε, νέες ε, διευθετήσεις στην αγορά, να πιέσουμε, αν θέλετε, με σωστό τρόπο τους παραγωγούς, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι τελικά δεν ενεργοποιούνται. Είναι επίσης πολύ σημαντικό η παραγωγή εκτός Ευρώπης να τύχουν προστασίας. Ή δεν μπορούμε εδώ να απομονωθούμε. Παραδείγματο χάρη, προστατεύουμε τους παραγωγούς οπωροκυπευτικών στην Ισπανία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να παρακαμφθεί και να παρεκκλίνει, αν θέλετε, ο εφοδιασμός σε μία άλλη περιοχή, στην ε, άλλη πλευρά της Μεσογείου, εκεί που δεν προστατεύονται οι παραγωγοί και ο εφοδιασμός, η προμήθεια να γίνει κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε και τους παραγωγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας να στηρίξουμε την ανάπτυξη, να στηρίξουμε την συνεργασία. Επαναλαμβάνω και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προστατεύσουμε τους παραγωγούς που βρίσκονται εκτός της Ευρώπης. Ο κύριος Τσούλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω όταν μιλάμε για θέμετες πρακτικές, ειδικότερα στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ένα σαφή ορισμό της αθέμητης εμπορικής πρακτικής. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αφήνει να εννοηθεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μέρων. Δεν ε, υπάρχουν πρακτικέ αθέμητε. Αυτό όμω δεν είναι αληθέ. Έχουμε πολλές φορές ε, ανισορροπία εξουσιών ε, και ο πιο αδύναμος ε, δέχεται την πρακτική και σιωπά. Η οδηγία λοιπόν σίγουρα κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι απολύτως σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα καταγγελίας των ε, πρακτικών ε, από τρίτους, από εξωτερικούς που να μην συμμετέχουν άμεσα στις ε, δυναμικές αυτές της αγοράς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε οι αγορές να γίνουν πιο διαφανείς και πιο δίκες και για τους καταναλωτές. Και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μας, υποστηρίζουμε αυτού του είδους την προσέγγιση. Αναμένω λοιπόν ότι και η Κομισιόν την κατάλληλη στιγμή θα προσθέσει και αυτή την πτυχή που έλειπε από την πρόταση της. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη προς το καλεσμένο μας και τους συναδέλφους αλλά συμπίπτει τη συνεδρίασή μας με τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΚΟ που συστάται το Brexit. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να είμαι εδώ από την αρχή. Α, μας το παράδειγμα των παγωτών Χονάκη. Ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Γιατί είπατε ε, ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα υποφεληθούν οι γεωργοί. Γιατί αν ισχύει αυτό, γιατί ισχύει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία ώστε να υποφεληθούν και οι παραγωγοί, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι. Μπορεί να κατάλαβα τελείως λάθος την πρόταση, αλλά όταν βλέπω τη διαφάνειά σας ε, που αναφέρει τους μικρούς γεωργούς, Εδώ μιλούμε για οργούς. Αν εσείς ε, αναφέρεστε σε μικρούς γεωργούς, τι είναι ακριβώς εννοείτε, πώς θα περιγράφετε ένα μικρό γεωργό, άντρα ή γυναίκα. Επίσης, ε, Έχουμε διαφορετικά κρατημέλη με πολύ διαφορετικές πραγματικότητες ε, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή. Θα πρέπει όμως η νομοθεσία μας, όποια και αν εγκρίνουμε, να εφαρμοστεί επιτέλους, γιατί έχουμε ακούσει αυτές τις υποσχέσεις, αλλά δεν έχουμε ακόμη δει από την νομοθεσία. Και θέλουμε και καλή επιχειρηματολογία. Αλλά πώς έχω ακούσει μέχρι στιγμής και από αυτά που έχω μάθει από την παρουσίασή σας, όπως με ενημέρωσε η βοηθός, δεν υπάρχει αυτή η βάση, μια διάστη επιχειρηματολογία. Και αν ακολουθήσουμε την αρχική πρόταση, ποιο είναι το ποσοστό της αγοράς που επηρεάζεται. Έγινε Κατανοητή η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαζό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας πω ότι πραγματικά έχω μείνει άναυδος από το κατά πόσο είναι απόντες εδώ τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Εξίσου με σοκάρει αυτό όσο και οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πρόκειται για κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους εμπλεκόμενους, κάτι το καθοριστικό θα έλεγα. Στις τροπολογίες μας θελήσαμε να διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται προστασία για τους μικρούς, μεσαίους και μεγάλους ε, σημαντικούς γεωργούς, γιατί φυσικά και οποιοδήποτε αγρότης είναι πάντα μικρότερος και πιο αδύναμος από μια ε, μεγάλη αλυσίδα ε, αγοραστών και φυσικά και η αγροδιατροφική βιομηχανία, οι κεντρικές αγορές έχουν πάντα περισσότερες δυνατότητες, περισσότερο προσωπικό και θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι γεωργοί μας έχουν υποστεί ασφυκτική πίεση και είναι εξαιρετικά σημαντικές οι συνέπειες ε, για την παραγωγή αυτών των αθέμητων πρακτικών. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα η Ουκρανία ή η η Ισία έχουν υποφεληθεί από μια εξαιρετικά ευνοϊκή πολιτική. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες εντός και εκτός Ευρώπης λιώνουν και εμποδίζουν τους αγρότες μας να διαπρέψουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι όλοι μιλούν διπλωματικά. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η πραγματικότητα πραγματικά σήμερα βρίσκεται πολύ μακριά από την πραγματικότητα, από την πραγματικότητα που ζουν και βιώνουν καθημερινά οι αγρότες μας. Σας παρακαλώ πολύ, Μπορείτε να μου πείτε κάποιος που έχει 5 εκτάρια, 20 εκτάρια, 25 εκτάρια, τι βιώνει, ποια είναι η πραγματικότητά του καθημερινά, τι αντιμετωπίζει όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με την μεγάλη ε, διαπραγματευτική δύναμη και τα όπλα που διαθέτουν σήμερα οι μεγάλοι αγοραστές. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφάνεια σε αυτές τις εμπορικές πρακτικές. Υπάρχουν τέλη και σημαντικά βάρη επί του κάθε αγρότη σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομία της αγοράς, θα μου απαντήσετε, ναι, η οικονομία της αγοράς όμως πολλές φορές είναι απαραίτητη για να ρυθμίσει κάποια πράγματα και αυτό το βλέπουμε με τη φορολογία. Ο ανταγωνισμός σήμερα είναι κάτι που σίγουρα πολλές φορές ρυθμίζει καλύτερα ίσως από τη δική μας νομοθεσία. Θα πρέπει να δούμε τα μεγάλα, οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες πολυεθνικές, πώς ακριβώς διαπραγματεύονται. Σήμερα με αυτά που προτείνουμε δεν λύνουμε απολύτως κανένα πρόγραμμα μεταξύ των παραγωγών και των μεγάλων πολυεθνικών που διαπραγματεύονται τα προϊόντα τους. Οι αλυσίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον αυτό ισχύει στην Γερμανία, όταν διαπραγματεύονται με τις ενώσεις παραγωγών, με τους συνεταιρισμούς παραγωγών. Βεβαίως και λαμβάνουν υπόψη τους ε, την πραγματική τιμή, το κόστος, αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και πάρα πολλοί ενδιάμεσοι μεταποιητές. Σήμερα θα πρέπει ένα κοινοβούλιο, ένας νομοθέτης να μπορεί να αποφασίσει για τους όρους και τις προϋποθέσεις και όχι ένας όμιλο σούπερ μάρκετ ή μια πολυεθνική. Και ο σκοπός μας εδώ είναι πραγματικά να προστατεύσουμε τους γεωργούς. Ευχαριστώ κύριος Άγγλιο. Ευχαριστώ. Εδώ μιλούμε για θέμετες εμπορικές πρακτικές και τη σχετική νομοθεσία. Ο κύριος Βαλέτη, ο δόκτωρ Βαλέτη, ο καθηγητής Βαλέτη, θέλω να σας προσβάλλω, δεν αναφέρω στο τίτλο, ε, είπε ότι πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση όταν κατεβούμε λίγο κάτω από την επιφάνεια. Και μάλιστα μερικοί παραγωγοί θέλουν προώθηση, γιατί έχουν ένα καινούργιο προϊόν και μόνο με κάποια έστω και βραχυπρόθεσμη επιδότηση μπορεί να το προωθήσουν. Μάλιστα έχω υποστεί πιέσεις από λόμπι και λενοπολιτών και μεταποιητών. Οι λενοπολιτές λένε ότι γίνονται τα θύματα, ε, γίνονται πολλά, ε, κερδοσκοπούν οι μεταποιητές και τα θύματα είναι ίδια. Ενώ οι μεταποιητές από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι αν προσπαθήσουν να διεκδικήσουν υψηλότερη τιμή για το προϊόν, το σούπερ μάρκετ θα τους ξεγράψει από το κατάλογο. Και ξέρουν ε, τα σούπερ μάρκετ ότι δεν έχουν πουθενά άλλο να αποταθούν οι μεταποιητές. Οπότε και οι μεταποιητές και οι λιανοπολιτές ε, ε, μου ασκούν πιέσεις με τα δικά τους επιχειρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαβεβαίωσε εδώ στην Επιτροπή Άγκρη ότι η προτινόμενη νομοθεσία δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες ε, του δικού μας ε, συνηγόρου των σούπερ μάρκετ, όπως λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά τι θα γίνει με το Υπουργείο Γεωργίας που θα χρειαστεί να αυξήσει το προσωπικό του συγκεκριμένου διαμεσολαβητή από 2 σε 50 άτομα αυτού του διαμεσολαβητή του σούπερ μάρκετ γιατί θα πρέπει συνέχεια ε, αυτή η αρμόδια διαμεσολαβήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο να ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζονται τέτοιε αθέμητε πρακτικέ ή όχι, ελέγχοντα τα σούπερ μάρκετ. Επίση, ε, τι γίνεται με αυτέ τι μονομερεί συμβάσει, όπου ο λιανοπολιτή ε, μπορεί να ρίξει τον παραγωγό πολύ γρήγορα και τελευταία στιγμή, ενώ ο προμηθευτής θα πρέπει να ακολουθεί μια πολύ μακροχρόνια προθεσμία προειδοποίησης. Αυτό είναι άδικο. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά Βαλέτη, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι το... η νομοθεσία αυτή είναι απαραίτητη και την περιμένουμε και τη ζητούμε εδώ και πολύ καιρό. Μιλούμε για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που είναι βαθιά ριζωμένες. Υπάρχουν ακόμη και εταιρείε παροχή συμβουλών που δίνουν συμβουλές για το πώς θα αποφευχθούν από τους ενδιαφερόμενους οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Θέλουμε επιτέλους μια νομοθετική πράξη που θα βάλει λίγη τάξη στην αλυσίδα εφοδιασμού εμβιορικών προϊόντων και τροφίμων. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε στη μοίρα του του εμπλεκόμενου να αντιμετωπίζουν από μόνοι τους τι εμπορικές, εμπορικέ πρακτικέ. εμπορικές πρακτικές. Επίσης, οι προμηθευτέ πρώτων υλών στη Γεωργία έχουν πολύ ασθενή διαπραγματευτική θέση και ελάχιστη διαπραγματευτική δύναμη και έχουν, ε, είναι στριμωγμένοι στον τοίχο. Και ξαφνικά ε, έχει ε, μειωθεί το βούτυρο. Αν δεν κάνουμε τίποτα, την αύριο δεν θα έχουμε ούτε λουκάνικα στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε κάτι περαιτέρω των άμεσων ενισχύσεων. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε την αγορά για να μην έχουμε λήψεις ε, γεωργικών προϊόντων. Επίσης, μιλούμε για ελεύθερη αγορά. Αν όμως δεν ρυθμίσουμε τις τιμές, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τουλάχιστον τις σχέσεις μεταξύ των κρίκο της αλυσίδα, ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να απολούν τα προϊόντα τους, στα προϊόντα τους αξιοπρεπείς τιμές και να μπορούν να επιβιώνουν χάρη στη δραστηριότητα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ένα ελάχιστο όριο τιμών. Και κάτι επιπλέον, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε γιατί έχουμε τόσο τεράστιες διαφορές στην ενιαία αγορά. Γιατί έχουμε μια ενιαία αγορά, αλλά 28 χώρες μέλη. Και οι τιμές γάλακτος, για παράδειγμα, έχουν ε, τεράστιες διαφορές. Μερικές φορές έχουμε τριπλάσιες, τετραπλάσιες τιμές στο λίτρο γάλακτος στις διάφορες χώρες. Επίσης έχουμε παραγωγούς, έχουμε προμηθευ... μεταποιητές, έχουμε αγοραστές και πολιτές. Όλοι αυτοί είναι κρίκοι της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα πρέπει λοιπόν η νομοθετική αυτή πρόταση να είναι όσο πιο οριθετημένη γίνεται για να έχει πραγματικό και θετικό αντίκτυπο. Πόσο ο κύριος Ντόρφμαν. Τάνκε. Ευχαριστώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε, ιδιαίτερα όσον αφορά την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Πρέπει να σας πω ότι κάπως ξεπνιάστηκα. Εδώ κάτω από το κτίριο αυτό υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να πάτε και να δείτε ποια είναι τα προϊόντα, πόσα είναι τα προϊόντα αυτά που κατευθείαν ε, έρχονται και είναι προϊόντα ντελές ή άλλων μεγάλων ομίλων. Μπορείτε να μην βρείτε πολλές, ε, αν θέλετε, προϊόντα από ποικιλίε που έρχονται κατευθείαν από τους παραγωγούς. Αλλά τελικά βλέπετε ότι η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ αυτών των μεγάλων σοπερμάρκετ, μεγάλων ε, ομίλων, και των παραγωγών ή των ενώσεών τα. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή όπου περίπου το 10% της παραγωγής μήλων ε, παράγονται εκεί. Και πρέπει να σας πω ότι τελικά η παραγωγή, όλη αυτή η παραγωγή περνάει από οργανώσεις παραγωγών, από συνεταιρισμούς και δύο τον αριθμό, καταλαβαίνετε, ότι δεν υπάρχει ο μικρός παραγωγός τον οποίο πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δυνατότητα να γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις με έναν τρόπο βάσει κανόνων. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είτε αγοράτε μήλα, είτε αγοράτε αχλα... αγοράζετε αχλάδια. Τι μπορεί να κάνει τελικά το σούπερ μάρκετ που τα πουλάει. Είτε γίνεται κάτι αν θέλετε επίτηδες για να πιέσουν τον παραγωγό, είτε πρέπει να μιλήσουμε για τους κανόνες της αγοράς, την οικονομία της αγοράς και να το δούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Ντόρφμαν. Θεωρείτε, κύριε Βαλέτη, ότι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές στις μεταπητικές εταιρείε ε, επηρεάζουν το σύνολο της αλυσίδας ε, εφοδιασμού, ακόμη και τον παραγωγό ε, που προμηθεύει τους μεταπητές. Γιατί αν ακολουθήσουμε τη δική σας λογική, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται. Κάποιες χώρες ήδη έχουν νομοθεσία που καλύπτει το σύνολο των πρακτικών, των εμπορικών πρακτικών. Οπότε, αν δεν προστατεύσουμε τους μεσάζοντες, σε τελική ανάλυση ο παραγωγός της πρώτης ύλη θα γίνει το θύμα αυτής της αλυσίδας λόγω της πίεσης που ασκείται πάνω του από το σύνολο των υπόλοιπων κρίκων της αλυσίδας. Και μάλιστα το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποδείξει στις αναλύσεις του ότι μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές που θα καλύπτει όλους τους προμηθευτές δεν θα έχει αποπληθωριστικό αποτέλεσμα στις τιμές λιανικής. Ερωτώ λοιπόν, γιατί ε, αντιμετωπίζετε διαφορετικά τη γεωργική παραγωγή σχέση με τις υπόλοιπες παραγωγές. Γιατί κάνετε αυτό το διαχωρισμό θεωρώ ότι η προσέγγιση της κυρίας Μαγκίνης και του καθηγητού Ντεκάστρο είναι πολύ ισορροπημένη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε στην αίθουσα καλεσμένους της κυρίας Αγγιλέρα, μια ομάδα γεωργών από την Ανδαλουσία. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και παρακολουθείτε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ε, I'd like to welcome the two. I used to live... Εγώ είσαι εκεί για δύο μήνες, ήταν καταπληκτικά. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με μια από τις τροπολογίες και σε ποια λογική βασίζεται όσον αφορά τον ορισμό της οικονομικής εξάρτησης ως 20% και προτείνω να το αλλάξουμε σε σημαντική εξάρτηση και έχει γίνει πρόταση να τα αλλάξει σημαντική εξάρτηση. Αναρωτιέμαι, το σημαντικό σημαίνει διαφορετικό για, κάποιο, για τον καθένα. Δεν αποδυναμώνουμε εδώ, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Γιατί οδηγία και αντικανονισμό και, και όχι κανονισμό, για ποιο λόγο επιλέξετε οδηγία έχουμε περίπου 20 χώρες που έχουν σχετική νομοθεσία και μέτρα για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ο κύριος Χόισλινγκ. Πιστεύω, και το είπαν και άλλοι σημαντικοί συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής και θα πρέπει να δούμε τελικά ποιον θέλουμε να βοηθήσουμε, ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε. Και γι' αυτό και η συζήτηση μικρή-μεγάλη παραγωγή δεν είναι αδικαιολόγητη. Πιστεύω ότι εδώ στο κείμενο δεν αναφερόμαστε μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες γεωργών. Βλέπω παραδείγματος χάρη ότι αναφέρομαι σε κάποιους συνεταιρισμούς Αναφερόμαστε σε συνεταιρισμού μικροπαραγωγών, σε μικρομεσαίες επιχείρησεις. Δεν ξέρω, η Επιτροπή κάπω θα πρέπει να οριοθετήσει τις κατηγορίες αυτών που προστατεύουμε. Υπάρχουν συνεταιρισμοί και συνεταιρισμοί. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ και των παραγωγών και των ενώσεων παραγωγών και γι' αυτό και προτείνω να γίνουν πιο συγκεκριμένοι και σαφείς οι ορισμοί. Τελικά, αυτούς που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι η παραγωγή. Και δεν έχω την εντύπωση δικά που στο κείμενο με σαφήνεια το αναφέρουμε αυτό. Και ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω. Και αναφέρομαι στον κύριο Ντες. Το θέμα που ανέφερες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το θέμα της διαπραγμάτευσης και μεταξύ ποιου γίνεται και το θέμα του πώς επιλέγουμε κάποια προϊόντα. Ξέρετε πολύ καλά πώς επιλέγω τα προϊόντα, πολλές φορές αποκλείονται προϊόντα, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να ασκηθεί η πίεση των παραγωγών για να χαμηλώσουν οι τιμές. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η εμπορική πολιτική. Δεν ε, θα εμποδίσουμε και θα απαγορεύσουμε εμείς σε μια επιχείρηση να θεσπίσει τα δικά της κριτήρια επιλογής. Το θέμα του προστατευτισμού είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε επάπειρον και δεν μπορούμε βεβαίως εδώ να πούμε σε μια επιχείρηση ότι μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε με όποιο τρόπο θέλετε. Και θα πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα, παραδείγματος χάρη, στους παραγωγούς μιας περιοχής κατά προτεραιότητα να αγοράζονται τα προϊόντα της περιοχής, της περιφέρειας. Κάποια κριτήρια δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που έφτασα καθυστερημένα, αλλά ήμουν στην Επιτροπή Ελίας. είχαμε και ψηφοφορίες και έχασα δυστυχώς την παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, παρουσίαση της έκθεσης του κ. Ντακάστρο. Πάντως, ε, μια και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, θα ήθελα να πω ότι η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Εξαιρετικά σημαντική και χαίρομαι που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια νομοθετική πρόταση για να τη συζητήσουμε. Επίσης, θεωρώ πολύ σωστό, α, πολύ σωστές είναι οι προτάσεις α, της έκθεσης Δεκάστρο, παρόλο που θεωρώ ότι και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή. Το πεδίο εφαρμογή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Θα πρέπει δηλαδή να προστατεύσουμε τους γεωργούς και όλους τους κρίκους αλυσίδες από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Συγγνώμη για το κινητό μου. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, αλλά το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε του γεωργού απέναντι στι πρακτικέ αυτέ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το κύριο μέλημα τη οδηγία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο από οποιαδήποτε άλλη πτυχή τη κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει επίση να διορθώσουμε τι πολύ χαμηλέ τιμέ που λαμβάνουν για τα προϊόντα του Γεωργοί. Αν δεν διορθώσουμε αυτέ τι αθέμετε εμπορικέ πρακτικέ στην αλυσίδα εφοδιασμού, δεν πρόκειται να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη σε αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Και η εμπειρία που έχουμε ε, είναι κατά τις παρέμβαση ε, στι τιμέ καταναλωτή. Έχω υποβάλει μια τροπολογία που θα ήθελα να γίνει δεκτή. Πρόκειται για πωλήσει ε, με ζημιά, σε τιμές κάτω του κόστους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, η πώληση ε, με ζημία. Είναι μια αθέμητη εμπορική πρακτική, κατά τη γνώμη μου, και αυτή η πρακτική της πώληση σε τιμές κάτω του κόστους, με ζημία δηλαδή. Είναι πολύ σωστή λοιπόν και εύστοχη η πρόταση αυτή. Θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση και να δούμε τι ε, συνέπειες έχει μία πρακτική πωλήσεων σε τιμή κάτω του κόστου, σε τιμή όπου με βγαίνει ζημιωμένος ο παραγωγός. Σίγουρα είναι και αυτό αθέμητη εμπορική πρακτική. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή, να το διευρύνουμε για να έχουμε μια καλή νομοθεσία. Οποιαδήποτε αθέμητη εμπορική πρακτική είναι κακή, είτε αν γίνεται προ τα πάνω είτε αν γίνεται προ τα κάτω. Ποτέ όμω δεν γίνεται προ τα πάνω. Συνήθω γίνεται προ τα κάτω. Δηλαδή πιέζει, συμπιέζει του γεωργού και πειράζει το γεωργικό εισόδημα. Ενώ οι καταναλωτέ ουδέποτε δεν, δεν ευνοούνται από μια αθέμητη εμπορική πρακτική. Αυτοί που ευνοούνται είναι κυρίω στα σούπερ μάρκετ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των αγορητών από την Ομίγυρη, λέει ο πρόεδρο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να απαντήσει. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Δεκάστρο. Πρώτα όμω τον κύριο Βαλέτη. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και φάνηκε από το ζωηρό ενδιαφέρον και το πάθος με το οποίο το σχολιάσατε και θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την ομάδα γεωργών από την Ανταλουσία που κατάλαβαν ότι η συζήτηση που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορά την πραγματικότητα στην Ευρώπη και τα πραγματικά τους προβλήματα. υπάρχουν διαφορετικές πτυχές και διαφορετικές πραγματικότητες και προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή λύση για τα κράτη-μέλη και μερικές φορές ε, το να προσπαθεί κανείς να προβάλλει τα εθνικά του προβλήματα σε ολόκληρη την Ένωση οδηγεί σε δυσκολίες. Και όταν προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των πρακτικών που έχουμε χαρακτηρίσει κακές, αθέμητες, δεν θεωρούμε ότι είναι οι μόνες, οι μοναδικές. Απλώς δεν είναι τόσο παρούσες οι πιο γενικευμένες, εκτός από από μια χώρα ώστε να ε, δικαιολογούν διαφορετική ε, μεταχείριση ή να είναι εκτός του καταλόγου. Οπότε ε, με την πρόταση αυτή δίνουμε την εξουσία και την ισχύ στα κράτη-μέλη που έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ακόμη πιο φιλόδοξες και πιο αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις αν θεωρούν ότι κάποιες αθέμητες πρακτικές που είναι παρούσες στη χώρα τους επηρεάζουν τους παραγωγούς. Ε, δεν μπορεί, δεν μπορεί λοιπόν μια χώρα να είναι, λιγότερο, να είναι πιο επικής, να είναι λιγότερο αυστηρή, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι πιο αυστηρή στα μέτρα της. Επίσης, δεν καταργούμε καμία νομοθεσία ή δεν αποσυρώμαστε από καμία νομοθεσία. Απλώς προσπαθούμε να βρούμε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Δεν υπάρχει μια μέση ευρωπαϊκή χώρα. Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων προοπτικών και των διαφόρων πραγματικότητων στα κράτη-μέλη. Αυτά ως γενική εισαγωγή. Πάντως είναι σημαντικό να το επισημάνω. Κάτι άλλο κοινό, ένα άλλο κοινό στοιχείο που ανέκυψε από τη συζήτηση είναι ότι φαίνεται ότι ενστικτοδός θέλετε να εφαρμόζονται κάποια νομοθετικά μέτρα στη σχέση μεταξύ μεγάλων παικτών, μεγάλων παραγωγών, μεγάλων μεταπίτων, μεγάλων πολιτών, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Όχι ότι είμαι καταρχήν κατά μια τέτοια πρόταση, αλλά στην πράξη μπορούν να γίνουν πολλέ παρακάμψει ε, και να έχουμε ανεπιθύμητε ε, ε, συνέπειε. Στη Τσεχία, για παράδειγμα, η Coca-Cola, που είναι γνωστό από, είναι πολυεθνική και ανήκει στου πολιτέ, κατάφερε να χρησιμοποιήσει και μάλιστα να κάνει κατάχρηση του εθνικού συστήματος αθέμητων εμπορικών πρακτικών για να εμποδίσει ε, ή να επηρεάσει την διαπραγματευτική ισχύ των αγοραστών στην αγορά που έχουν το 10% μερίδιο της ε, αγοράς. Αυτό είναι καλό. Θέλετε να επιτρέψετε τέτοιου είδους δυνατότητα, τέτοιου είδους ε, περιθώρια λιγμών για τις πολυεθνικές. Όχι, προσοχή λοιπόν. Θα πρέπει να δούμε πόσα αντίθετα παραδείγματα έχουμε. Τώρα, έρχομαι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μερικές θα μπορέσω να τι απαντήσω, άλλες δεν θα μπορέσω γιατί είμαι ένα απλό οικονομολόγος. Αν θα πρέπει να είναι οδηγία ή κανονισμό δεν αναπόκειται σε μένα να το κρίνω. Επίση, και εγώ βλέπω μερικά πολύ σημαντικά πράγματα. Αναφέρθηκε το Μαρόκο, για παράδειγμα, από την κυρία Χόιμπουχ, από τον κύριο Χόισλινγκ. Και λοιπόν, αν προφέρω λάθος τα ονόματά σας. Θα, μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, μακάρι. Και σίγουρα μας προβληματίζουν ε, οι Μαροκινοί Γεωργοί, γιατί θέλουμε ε, γεωργική ανάπτυξη και για αυτούς. Αλλά αυτό είναι μια νομική πτυχή που δεν μπορώ να τη σχολιάσω εγώ, γιατί όπως είπα είμαι οικονομολόγος. Μια μερική απάντηση στην ερώτηση του κυρίου Δεκάστρο ή στο σχόλιο του κυρίου Δεκάστρο. Εμείς στην ε, μελέτη μας δεν λέμε ότι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές ελληνικής. Εμείς στην μελέτη μας θέλουμε να δούμε πώς οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές επηρεάσουν τους γεωργούς. Ποια είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπο γεωργού. Και αυτή, αυτό είναι το σημείο αφετηρία. Θα πρέπει να υποφελούνται από τι εμπορικέ πρακτικέ οι γεωργοί πρώτα απ' όλα. Επίση υπάρχει αυτή η κατακόρυφη πτυχή της αλυσίδα. Αλλά σε τελική ανάλυση θέλουμε η γεωργή, η παραγωγή να είναι κερδισμένη της συζήτηση. Αυτοί να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Και η άμεση, ο άμεσος δεσμός μεταξύ των παραγωγών και αυτών των αγοραστών είναι εμφανής. Αλλά υπάρχουν κάποια άδειλα σημεία και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτές τις έμεσες ε, σχέσεις. Επίση, ε, ο αντίκτυπο των εμπορικών πρακτικών στι τιμέ πώληση δεν ήταν το αντικείμενο της ε, μελέτη επιπτώσεων, της μελέτη αντικτύπου. Τώρα, για το θεμητό και το αθέμητο, ε, η έννοια της δικαιοσύνη του θεμητού, είναι κάτι που με αγγίζει και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος αυτό, αλλά θα πρέπει να το δούμε και λειτουργικά, γιατί το δίκαιο και το θεμητό είναι μερικές φορές υποκειμενικό θέμα. Και σίγουρα σε πολλές συζητήσεις θα προταχθούν ε, οικονομικά συμφέροντα. Και πολλές φορές αυτά είναι στο παρασκήνιο και πολύ συχνά μεγάλοι αγοραστές και πολιτές με μεγάλη αγοραστική ισχύ θα έχουν την επιρροή να πούν ότι όχι δεν είναι δίκαιο. Και εσείς μπορείτε να προσλάβετε κάποιον άλλον οικονομολόγο που δεν θα έχει το ίδιο δικαίω αίσθημα και θα κρίνει διαφορετικά το δίκαιο ή το θεμητό. Οπότε είναι σημαντικό η πρόταση να είναι ρεαλιστική, πραγματιστική και να δούμε και τι εναλλακτικέ υπάρχουν. Να δούμε οι εναλλακτικέ λύσει ε, μπορούν να εφαρμοστούν, ε, θα είναι εύκολα εφαρμόσιμες από τα κράτη-μέλη χωρί να απαιτούν πολλού πόρου. Είναι εφικτά τα μέτρα θα πρέπει αυτά τα φίλτρα λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε τις προτάσεις και τα μέτρα. Ο κύριος Φλανάγκαν μίλησε για την οικονομική εξάρτηση. Η οικονομική εξάρτηση είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε ε, ως οικονομολόγοι, αλλά απαιτεί πολλούς πόρους και εγώ καθημερινά προσπαθώ να βρω την αγοραστική ισχύ, τι ε, αγορέ, αλλά έχουμε πολλέ συγχωνεύσει το χρόνο, οπότε μπορούν να έρθουν οι παίκτε και να πείτε ε, είναι παγκόσμια αγορά, έχουμε ανταγωνισμό παντού και για να κρίνουμε κάθε φορά την κάθε συγχώνευση θα χρειαζόμαστε μεγάλο προσωπικό και η Γενική Διαθήση Ανταγωνισμού έχει αρκετούς πόρους αλλά έχει και τεράστιο και δύσκολο έργο και αν κάθε κράτος θα πρέπει περιπτωσιολογικά να κρίνει τι εστί η οικονομική εξάρτηση και αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί ίσως δεν μας οδηγήσει πουθενά μια τέτοια άγουσα. Έγιναν κάποιες απόπειρες από ό,τι ξέρω στη Γερμανία έγιναν κάποιες προτάσεις για τον ορισμό της οικονομικής εξάρτησης και η Κύπρος έκανε κάτι τέτοια, κάποιες τέτοιες προσπάθειες, αλλά η εφαρμογή είναι μηδαμινή. γιατί στο 2016 είχαμε μία περίπτωση με βάση την οικονομική εξάρτηση. Στην Κύπρο καμία τέτοια υπόθεση δεν είχαμε, γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τόσο αφηρημένες έννοιες όπως τις οικονομικές εξάρτησεις. Τώρα, γιατί αναφέρομαι στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, Γιατί είναι σαφώ προσδιορισμένε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μικρομεσαία είναι μια επιχείρηση που έχει μέχρι 250 υπαλλήλου και μέχρι 50 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Αυτό προσδιορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ομοιογενέ, ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη-μέλη τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Αν τώρα μια χώρα θέλει να ορίσει τη μικρομεσαία επιχείρηση σε επιχείρηση που έχει μέχρι 500 εργαζομένους ε, λόγω της ε, εθνικής πραγματικότητας, ε, δεν αποκλείεται. Μπορεί κανείς να είναι πιο αυστηρός. Επίσης, η κυρία Μακιντάιρ αναφέρθηκε στην ειδική διαμεσολαβήτρια που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο κύριος Άγγινου το ίδιο έκανε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιους διαμεσολαβητές αλλά όπω είπε ο κ. Σάγνιου, χρειάζεται μεγάλο προσωπικό. Θα πρέπει η διαμεσολαβήτρια να έχει το προσωπικό, του πόρου, τις γνώσεις για να κάνει κάτι τέτοιο, να ελέγχει τις αθέμητες εμπορικέ πρακτικές και θα πρέπει να είναι και ευχριστό και εφαρμόσιμο, εφικτό στην πράξη. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων, ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων. Δεν θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε με το στανιό κάτι. Ε, έχουμε κάτι τέτοιο στον ανταγωνισμό, γιατί έχουμε μακρά πείρα και μπορούμε ε, να εφαρμόσουμε τα θέματα ανταγωνισμού στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε ό,τι αφορά τι αθέμετε εμπορικέ πρακτικέ, τα κρατη μέρη έχουν πολύ περισσότερη εμπειρία. Εμεί προτείνουμε απλώ ένα σημείο αφετηρία, αλλά εσεί μπορείτε να το προωθήσετε και να το, να το ξεπεράσετε. Κυρία Μαγκίνες, να προσδιορίσω το παράδειγμα που έδωσα με το παγωτό χωνάκι. Θα το ξαναπώ. Αν η Unilever ε, διαπραγματεύεται τους όρους ε, προμήθειας κορνέτο, παγωτό χωνάκι, άλλη μορφή παγωτού προς το σούπερ μάρκετ Carrefour, εντάξει, ας το κάνει. Όποιο έχει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ισχύ και ικανότητα θα ε, τα καταφέρει. Τώρα, αν όμως την καλύψουμε ε, με τις θέμα τις εμπορικές πρακτικές και πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη τιμή για το κορνέτο, το παγωτό χωνάκι, ε, το θέμα είναι ποιος θα υποφεληθεί. Ο Βέλγος παραγωγός γάλακτος θα υποφεληθεί αν το παγωτό χωνάκι είναι ακριβότερο. Είπαμε όχι. Αν όμως το σούπερ μάρκετ, ο Σαν, Καρφούρ, ε, αγοράσει απευθείας το γάλα από τον κτηνοτρόφο το βέλγο, τότε θα καλύπτεται από την πρόταση της οδηγίας. Όχι όμως αν η Unilever το αγοράζει, το προμηθεύει στη, στο σούπερ μάρκετ. Επίσης, αν η Unilever προσπαθήσει να μετακυλήσει κάτι ή να πει «Α, συγγνώμη, ο παραγός κάτι μου δίνει α, σε εντάλλαγμα, αλλά τελικά ε, λόγω των ειδικών όρων που επιβάλλει το σούπερ μάρκετ ΣΑΝ, μετακυλίω τη ζημιά μου στον παραγωγό, στο κτηνοτρόφο. Αυτός ο έμεσος, ε, αυτή, αυτός ο έμεσος αντίκτυπος καλύπτεται από την πρόταση για να αποφευθεί η μετακύληση της ζημιάς στον παραγωγό. Επίσης, ο κύριος Ντες, ο κύριος Ντόρφμαν έκαναν κάποια σχόλια. Ναι, όλοι, όλοι Ευρωπαίοι είμαστε. Έχετε δίκιο. Με κατηγορήσατε ως εθεροβάμωνα. Μου είπατε ότι είμαι εκτός πραγματικότητας. Ότι είμαι στον για γυάλινο πύργο του ακαδημαϊκού κύκλου του Πανεπιστημίου και δεν έχω καμία επαφή με την πραγματικότητα. Σίγουρα αυτό είπα και προηγουμένως. Εσείς είστε σε άμεση επαφή με την πραγματικότητα γιατί έχετε πληροφορίες από τους ψηφοφόρους σας, τους γεωργούς σας, οπότε η πραγματικότητα η δική σας είναι διαφορετική από τη δική μου. Γιατί έχετε σχέση με την ε, νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Και σίγουρα η Ευρώπη είναι μια κοινή βάση απλώς. Τα κράτη-μέλη προχωρούν πιο πέρα από τη βάση αυτή. Ο πρόεδρος μου επισημαίνει ότι εξαντλείται ο χρόνος μου και γι' αυτό θα βάλω εδώ τελεία, ευχαριστώντας σας για την προσοχή. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαλέτη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Δεκάστρο για να ολοκληρώσει μετά τη συζήτηση που έγινε για την έκθεσή του. Μπαίνουμε στην ουσία, Πρόεδρε. Ακούσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση του επικεφαλής ε, οικονομολόγου της ε, Γενικής Διευθύνσης Ανταγωνισμού και μπαίνουμε τώρα στην ουσία. Ήθελα να σας ανακοινώσω ότι πριν από λίγο η Επιτροπή ΙΜΚΟ ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της τροπολογίας της συμβιβαστικής που διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Σας ε, Υπενθυμίζω, συναδελφοί, 678 ήταν οι τροπολογίε ε, για αυτή την πρόταση οδηγία ε, για την καταπολέμηση των αθεμητών ε, εμπορικών πρακτικών. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους τους κοιόδης, όλους όσοι συνεργαστηκαν γιατί από τις 42 ε, συμβαστικές τροπολογίες 30 για τα άρθρα και 12 για τις ιδεολογικές σκέψεις έγινε ομαδική εργασία και πιστεύω ότι μπορώ να πω πως όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν επί αυτών των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχουμε μόνο μία εξαίρεση, όπως είπε η συνάδελφος η κυρία Κατάινεν, η Άλντε, η ομάδα Άλντε ε, αποστασιοποιείται από μια από αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά Κατά τα άλλα έχουν λάβει την έγκριση της πλειοψηφίας των ομάδων. Θέλω να ξαναυπενθυμίσω σε όλους πόσο σημαντικό είναι να εγκρίνουμε αυτή την οδηγία μέχρι τα τέλη της θητείας. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες. Το έχουμε δει και στη σχετική συζήτηση και στη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Δεν μπορούμε να κινδυνεύσουμε να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Γι' αυτό το λόγο εμείς αμέσως μετά από την ψήφο στην Ολομέλεια, σας υπενθυμίζω θα γίνει στην εβδομάδα του Στρασβούργου τη 22 Οκτωβρίου. Αμέσω μετά λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε αμέσω τους τριμερεί διαλογού. ήδη εκείνη τη βδομάδα ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε πολιτική συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω κάποια πραγματάκια, όχι πολλά για να μην μακρηγορήσω οι προσπάθειες για τις συμβαστικές τροπολογίες ε, ασχολήθηκαν και με ένα θέμα που αφορούσε τον ε, κατάλογο, τη λίστα των αθεμητών πρακτικών. 200 τροπολογίες είχαμε μόνο για αυτό, για το άρθρο 3. Εμείς προσπαθήσαμε με πολλές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, προσπαθήσαμε λοιπόν να διευκρινίσουμε τον όρο, τον ορισμό, συγγνώμη, στο βαθμό του δυνατού ώστε όπως ακούσαμε και εδώ στη συζήτηση, να δίνουμε και στα κράτη-μέλη την ευκαιρία να προσθέσουν κάτι περισσότερο σε αυτό. Και όπως είπαμε μπορούν. Παρ' όλα αυτά η πολιτική πίεση όλων των ομάδων και οι 200 αυτές ε, τροπολογίες μας οδήγησαν στο να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή των τεσσάρων λευκών όπως λέγονται ε, αθέμητων πρακτικών και των τεσσάρων ή Τις τέσσερις μαύρες τις ε, επεκτείναμε στα ε, γραπτά συμβόλαια μη υποχρεωτικά για όλους, προσοχή γιατί αυτό θα έχει δημιουργήσει αλλιώς προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη. Τα γραπτά συμβόλαια λοιπόν, τα έντυπα συμβόλαια, εφόσον ε, ζητηθούν από τον προμηθευτή, ο αγοραστής δεν μπορεί να, τα, να αρνηθεί να τα παράσχει, εφόσον τα ζητήσει ο προμηθευτής αν ο προμηθευτής τα ζητήσει υποχρεούται να τα δώσει να υπογράψει τέτοιε συμβάσει ο αγοραστή. Ε, εκεί έχουμε μια διεύρυνση και η δεύτερη διεύρυνση αφορά τον κίνδυνο της ε, κατάχρησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από πλευράς του αγοραστή. Ξέρετε ότι γίνει μια μεγάλη συζήτηση που εμείς δεν, έχουμε, δεν την έχουμε κάνει, αυτή την οδηγία για τα ιδιωτικά σήματα, τα private label. Ίσως θα ασχοληθούμε με αυτήν σε κάποιο άλλο νομοθέτημα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ορισμένοι αγοραστές είναι βρίσκονται, έχουν στη διάθεσή τους ευαίσθητες πληροφορίες ε, και θα πρέπει να ε, το προσέξουμε αυτό, ε, γιατί θα μπορούσαν να, να καταχραστούν αυτών των πληροφοριών. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνουμε τις πωλήσει κάτω του κόστους. Ζητήθηκε από πολλές αυτές, ομάδες αυτό, το θέμα αυτό είναι δύσκολο αντιλαμβανόμαστε, αλλά ως κοινοβούλιο στη συμβαστική ε, τροπολογία του κοινοβουλίου θα έχουμε συμπεριλάβει τις πωλήσει κάτω του κόστους. Και όπως είναι σαφές, ε, όπως ξέρουμε Εκκρεμεί μια απόφαση του δικαστηρίου για μια υπόθεση στην Ισπανία, για την νομοθεσία την Ισπανική. Ήταν μεγάλη πίεση και δεν μπορούσαμε λοιπόν να μην λάβουμε υπόψη αυτή τη σημαντική ε, ποσότητα, τον σημαντικό αριθμό ε, τροπολογιών για αυτό το σημείο. Ήθελα να σας πω ότι το παιχνίδι ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την ψήφο στην Ολομέλεια θα έχουμε τεράστια πίεση όλοι μας. Και εύχομαι να καταφέρουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε μια ισχυρή θέση για το Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν πιο ευρεία που θα μας επιτρέψει, θα μου επιτρέψει εμένα να πάω στους τριμερείς διαλόγους με μια θέση που, με την οποία να συμφωνούν όλοι στο βαθμό του δυνατού. Γιατί η δουλειά που έχουμε κάνει, όπως και η δουλειά που κάναμε για τον κανονισμό Omnibus, ε, συμπληρώνει όλη αυτή την πορεία ε, ενδυνάμωσης ε, των μικρών επιχειρηματιών ε, και των γεωργών μας ώστε να ενισχυθεί η θέση του σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά. Ελπίζω λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση να παίξουμε ένα καλό ομαδικό παιχνίδι. Εδώ κλείνω κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουν να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες συνάδελφοι, έχουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δεκάστρο. Η εκθέση του κυρίου ε, Ντεκάστρο περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και είναι πολύ σημαντικό να οριστικοποιήσουμε αυτό το έγγραφο και να το εγκρίνουμε πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Γιατί πραγματικά το περιμένουν πώς και πώς οι Ευρωπαίοι Γεωργοί, γιατί θέλουν μια τάξη στην Ευρωπαϊκή Αγορά και ξέρουμε πόσο καίγονται για το θέμα αυτό. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες συμβαστικές λύσεις και θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες, κάποιοι συμβιβασμοί. Επίσης, η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς είναι συνδεμένη επιτροπή. Η κυρία Μαγκίνης είναι σκιώδη συγκέντρια και παρακολουθεί το θέμα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Μαγκίνες εκ μέρους του κύριου Δεκάστρα και δεν χρειάζεται, να μπορούσε και ο να το κάνει. Δεν χρειάζεται να μεσολαβώ εγώ και να ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνες εκ μέρους του κυρίου Δεκάστρα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαγκίνες. Και παρακαλώ τον Κύριε Ντεκάστρο έρθει να με αντικαταστήσει. Thank Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ήξερα για την ε, αντικαταστήση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και να σχολιάσω την παρουσίαση της Επιτροπής. Αναφερόμαστε σε οικονομικά συμφέροντα, πολύ σημαντικά και φυσικά είναι μια συζήτηση η οποία έχει κρατήσει καιρό σε αυτή τη δική αυτού του κοινοβουλίου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ είναι κάτι που αν θέλετε, παρακολουθείτε με ιδιαίτερη προσοχή από αυτούς που θέλουν να αποτύχουμε, ελπίζουν να αποτύχουμε και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κοιτάει το θέμα αυτό υπό την προοπτική της βιώσιμης προστασίας και λειτουργίας της αγοράς αλλά και της αλυσίδας εφοδιασμού στο τομέα των τροφίμων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή για την συνενετική του στάση. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που ακόμα θα πρέπει να ξαναδούμε, να βρούμε και άλλους συμβιβασμούς. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα αν θέλουμε να ολοκληρωθεί η εργασία. Και φυσικά όσο πιο μεγάλη πίεση υπάρχει από τους λομπίστες, τόσο πιο αποφασισμένοι πρέπει να είμαστε και ακριβώς ε, επειδή υπάρχει ασάφεια και έλλειψη διαφάνειας, πρέπει εμείς να προσθέσουμε σαφείς κανόνες και διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρίν Κατάιναν. Και μετά ο Διευθυντής Μέγκελ ήθελα να, σας δώσω το, δώσω το λόγο πριν τελειώσουμε. Παρακαλώ, Μάριν. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις για την πάρα πολύ αποτελεσματική και επικοδομητική εργασία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η οδηγία αυτή είναι κάτι που το επεξεργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Okay. Okay. Δεν ακούγαμε. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, προετοιμάζαμε αυτή την οδηγία εδώ και πολύ καιρό και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό το ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ θα περάσει κι άλλος χρόνος, αλλά αυτή είναι η διαδικασία και αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το αντικείμενο αυτής της οδηγίας. Μιλάμε για τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, για αλυσίδα εφοδιασμού και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίσουμε το νομοθετικό έργο που γίνεται στα κράτη-μέλη. Την ίδια ώρα στηρίζουμε τις περιοχές αυτές, τους παραγωγούς αυτούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους κρίκους αυτής της αλυσίας. Και όταν ε, υπάρχουν υπόνοιες ε, ή προκύπτουν πραγματικά αθέμητες πρακτικές, θα πρέπει να αποδείξουν την μη ύπαρξή τους τα μεγάλα λόμπι, οι μεγάλοι όμιλοι και οι πολυεθνικές. Ο παραγωγός έχει δικαίωμα σε γραπτή σύμβαση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθεί στο κείμενο και ελπίζω ότι θα επιταχυνθεί και η διαδικασία του τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή κύριο Μάγκελ για να κλείσουμε αυτό το σημείο. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα παρατείνω υπερβολικά τη συζήτηση. Θα ήθελα να καλύψω όμως ορισμένα σημεία τα οποία δεν κάλυψε ο κ. Βαλέτη. Για πολύ καλή αιτία σχετίζονται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων και για ποιο λόγο αποφασίσαμε οδηγία. Σε αυτή την ερώτηση θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα γιατί οδηγία και όχι κανονισμό, διότι εδώ ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία αφορούν το αστικό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Ασχολούμαστε με μια κατάσταση που ήδη καλύπτεται από την Εθνική Νομοθεσία σε 20 κράτη-μέλη. Υπό τέτοιε συνθήκε δεν θα ήταν καλό να δημιουργήσουμε ένα κανονισμό ο οποίο θα παρενέβαινε άμεσα στο νομικό καθεστώ πολλών κρατών μελών και που ενδεχομένω ε, θα υπερίσχε τη εθνική νομοθεσία με τρόπο ανέφικτο, μη εφαρμόσιμο τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, δημιουργούμε τους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να τα μεταφέρουν αρμονικά στη δική τους νομοθεσία ώστε να λειτουργούν χωρίς τριβές, χωρίς επικαλύψεις και χωρίς όλες τις δυσκολίες που θα είχαμε κανονικά σε περίπτωση κανονισμού. Γι' αυτό το λόγο εδώ θεωρούσαμε ότι ήταν πιο λογικό να έχουμε μια οδηγία. Το πρώτο θέμα που μας αφορά εδώ επίσης ήταν και η νομική βάση, το 40 παράγραφος 2 που σε συντονισμό με το 39 άρθρο τη ε, ε, Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει του κύριου στόχου τη κοινή γεωργική πολιτική. Να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε το εισόδημα των αγροτών. Αυτό είναι. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε λοιπόν από την εισοδηματική κατάσταση των αγροτών στο πεδίο εφαρμογή, στο αντικείμενο του κειμένου, και είναι ακραία περίπτωση αυτή τη Unilever εναντίον Carrefour, τόσο πιο δύσκολο είναι να συσχετίσουμε αυτή την κατάσταση της πολυεθνικής με το εισόδημα του Γεωργού και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος της νομικής βάσης. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε λοιπόν τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος η νομική βάση να μην είναι επαρκής ώστε να καλυφθούν τα όσα θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι η πρόταση της Κομισιόν προσπαθεί να επιτύχει μια καλή ισορροπία και να βάλει κάτι μπροστά στον νομοθέτη το οποίο, αυτός να μπορεί να, το οποίο να μπορούμε να υπερασπιστούμε επαρκώς σε ένα δικαστήριο αν καταστεί αναγκαίο. Το δεύτερο που θέλω να πω ε, ε, σχετίζεται με μια προσθήκη που πρόκειται να γίνεται για τις πωλήσει με ζημία. Εμείς είχαμε προτείνει η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, να αφορά τις καταστάσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Εδώ δεν μιλάμε για μια αθέμητη πρακτική στο πλαίσιο της σχέσης αυτής. Μιλάμε για μια πρακτική που χρησιμοποιούν οι λιανοπολιτές ή οι πολιτές χονδρικοί σε σχέση με τους πελάτες τους. Δηλαδή, μιλάμε για τη σχέση μεταξύ ε, ε, λιανοπολιτή και πελάτη στο τέλος της ε, αλυσίδας. Οπότε πρέπει να ασχοληθούμε με αυτήν σε ένα άλλο πλαίσιο. Η άλλη ερώτηση που ανέφερε ο κ. Ροπέ φορούσε το γιατί έχουμε διαφορετικά επίπεδα τιμών σε διάφορα κράτη-μέλη και σε διάφορες περιοχές. Από την εμπειρία μας ο βασικός λόγος είναι η διαφορά μεταξύ ε, λιματικών και πλεονασματικών περιοχών. Στι πλεονασματικέ περιοχέ σχετικά οι τιμέ είναι χαμηλέ. Στι ελληματικέ περιοχέ είναι σχετικά υψηλέ οι τιμέ. Στι ελληματικέ περιοχέ αυτέ ε, έχουμε απομακρυσμένο χαρακτήρα ε, βρίσκονται μακριά από εκεί όπου πραγματοποιείται κυρίως παραγωγή, οπότε είναι μικρότερη η σχέση ε, από ότι γίνεται στις πλεονασματικές περιοχές. Υπάρχει διαφορά στο πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, στο πώς ε, διαχειρίζεται ο τομέας την αλυσίδα προμηθειών και όλα αυτά. Για παράδειγμα, έτσι έχουμε ότι ε, μια τιμή ε, λίτρου γάλακτος που δεν είναι ίδια σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ε, πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε ότι η πρόταση αυτή που έχετε μπροστά σας θα επέτρεπε στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν και αυστηρότερα μέτρα, αν το θεωρήσουν αναγκαίο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουν στα χέρια του τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν καταστάσει εντό τη επικράτειά του, ε, ενδεχομένω πολύ διαφορετικέ από ένα άλλο κράτο μέλο. Όσο περισσότερο μπούμε λοιπόν εμεί σε λεπτομέρειε, πιστεύω, τόσο λιγότερο αφήνουμε ελεύθερα τα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν πολύ στοχευμένα συγκεκριμένε υποθέσει ε, και περιπτώσει ε, εντό τη επικράτειά του. Γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι εδώ λογικά χρησιμοποιείται η έννοια τη ελάχιστη εναρμόνιση και πρέπει να διατηρηθεί και στο τελική έκβαση των συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας επικοδομητικά στην όλη διαδικασία μας τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε. Χαιρετίζουμε την Κομισιόν. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Μέγκελ και ευχαριστούμε και τον προσκεκλημάνο μας, τον επιφαλής οικονομολόγο της Κομισιόν, τον κύριο Βαλέτα, τον κύριο καθηγητά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 ε, για την κυρία Ρέτζη. Η συνάδελφός μα η Μαρία Καμπρίελα Ζωάνα είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο Μαρία Γκαμπριέλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία εντάσσεται στην πρόταση του νέου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027. Θα έχουμε κοινέ διατάξεις για τα 7 αυτά ταμεία με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως έχουμε μία βάση λειτουργίας για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία και μέσω της εναρμόνισης και τους κοινούς αυτούς ε, κανόνες και τις κοινέ διατάξεις οι δικαιούχοι θα ευνοηθούν και κυρίως στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Έτσι θα ενισχυθεί η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θεωρώ ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο και εναρμονισμένο πλαίσιο ανάπτυξης για όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις περιφέρειες των κρατών μέλων. Και θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών των κρατών μέλων. Και έτσι το νέο πλαίσιο θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της συνέχειας, της απλούστευσης και της ευελιξίας στη διαδικασία της εφαρμογής. Δυστυχώς όμως, μία καινοτομία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας είναι ότι στον κανονισμό αυτό δεν γίνεται πια λόγος για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ταμείο ξέρετε Ας μην ξεχνούμε όμως ότι τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδοτούν πολλούς αναπτυξιακούς στόχους και οι δικαιούχοι είναι πολύ άριθμοι. Μάλιστα τα κονδύλια αυτών των ταμείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες επενδύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό τα ταμεία αυτά και τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και Συνοχή να εμπίπτουν στο ίδιο πλαίσιο. Οπότε θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί η χρήση των κονδύλιων αυτών και να εξασφαλιστεί καλύτερη δυνατή συνέργεια μεταξύ τους. Είτε σε περιφερειακό λοιπόν, είτε σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί αυτό το ταμείο είναι που εγγυάται τη συνοχή, την κοινωνική συνοχή που είναι τόσο σημαντική, όχι μόνο για τις αγροτικές περιοχές, αλλά και για τις αστικές περιοχές. Αυτό είναι το πρωταρχικό επιχείρημα που συνηγορεί υπέρ της ε, παραμονής του Γεωργικού Ταμείου στον μελλοντικό κανονισμό περί κοινών διατάξεων, που καλύπτει τα άλλα 7 ταμεία. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές ζώνες, γιατί όλοι θέλουμε να γεφυρώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση των αγροτικών περιοχών, των επιχειρήσεών τους και να συμβάλλουμε στην καλύτερη ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοκομείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της μειώνει κατά 27% τα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό μας δυσαρεστεί ιδιαίτερος και το κατακρίναμε και στην γνωμοδότηση που υποβάλαμε στην Ολομένη και που εγκρίθεται. Αυτή η μείωση κατά 27% των περιφερειακών κονδυλίων είναι απαράδεκτη. Και δημιουργείται ένας αυξημένος κίνδυνος να μειωθεί περαιτέρω ο προϋπολογισμός των διαρθρωτικών ταμείων. Θα πρέπει λοιπόν ε, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο, Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξης να μεταχείριση μεταχείρισης με τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταμεία. Και ω μέλο και τη επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη, το συζήτησα με τους συναδέλφους και σας διαβεβαιώ ότι η πλειοψηφία των μελών τη ΡΕΓΚΙ συμφωνεί μαζί μου. Κατά την εκπόνηση των τροπολογιών προσπάθησα να σταθώ σε μία απλούστευση, δηλαδή να εξασφαλίσω την ευελιξία των διατάξεων που είναι παρόμοια με αυτή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό για την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτή είναι η πρότασή μου λοιπόν, να συμπεριληφθεί και το γεωργικό ταμείο στα, ταμεία και ο κατάλογος που υπάρχει στον κανονισμό για την ΚΑΠ να συμπεριληφθεί και στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνεί γιατί θεωρείται κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στη συγχώνευση των δύο πυλώνων της κοινή γεωρικής πολιτικής. Εγώ δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι με τις τροπολογίες μου δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα και μπορούν κάλλιστα οι διατάξεις αυτές περί κοινή γεωρικής πολιτικής να περιληφθούν στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Πιστεύω ότι κρατούμε ανοιχτέ ε, τις πόρτες και έχουμε και μία άμεση σύνδεση με το κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Γιατί λοιπόν να μην διαρευνήσουμε όλε τι εναλλακτικέ λύσει, Η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργικής πολιτική δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Δεν μπορούμε λοιπόν σήμερα να λάβουμε κάποιε οριστικέ αποφάσει και να αποκλείσουμε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής ανάπτυξη από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Κατά τη γνώμη μου, οριζόντιο αυτός κανονισμό περί κοινών διατάξεων έχει άμεση σχέση ε, με τον κανονισμό ο οριζόντιος κανονισμός έχει πολλά κοινά σημεία με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Και γι' αυτό με τις τροπολογίες μου διευκολύνεται αυτή η σχέση και συσφίγγονται οι δεσμοί μεταξύ των δύο κανονισμών και επιμένουμε στη συμπερίληψη του Γεωργικού Ταμείου στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Έτσι αποφεύγουμε την επικάλυψη των κανόνων και απλουστεύουμε το διοικητικό άχθος. Ταυτόχρονα επιτρέπουμε μια συνεκτική διαχείριση όλων των διαρθρωτικών ταμείων. Ξέρω ότι το ζήτημα είναι αρκετά λεπτό και ευαίσθητο, πάντως πιστεύω ε, ότι σε συνεργασία με τους και οδησηγητές θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Η 26η Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που λύγει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και με το ξεχνάτε αγαπητοί συνάδελφοι και περιμένω με ενδιαφέρον τη συνέχεια της συζήτησης. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ Ζωάννα. Κυρία Ζωάννα, τώρα θέλουν να μιλήσουν η κυρία Ρόπε και η κυρία Μαγκίνες. Και η κυρία Κύριε Ρόπε, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκφράσουμε την ε, δική μας θέση και να την υποβάλουμε στην Επιτροπή Ρέγκη. Εκείνοι θα αποφανθούν επί της ουσίας, θα επεξεργαστούν την ουσία. Φυσικά και χρειάζεται περισσότερη συνοχή. Συμφωνώ με την πρόταση ότι αυτό το μείον 10% είναι κάτι το απαράδεκτο. Το έχουμε εκφράσει εξάλλου και σε άλλα έγγραφα. Αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν 1,36% του 1% που συνεισφέρουν τώρα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να περικοπούν από αλλού τα κονδύλια της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Τι μήνυμα στέλνουμε. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε συνοχή σε αυτό το έγγραφο, όπως ακριβώς έχουμε εκφραστεί και τοποθετηθεί και αλλού. Πιστεύω επίσης ότι η συρρήκνωση και το πώς θα περικόψουν τα κράτη-μέλη κάποια από τα κονδύλια είναι κάτι που θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να έχει συνοχή. Οι ποσοστώσεις επίσης ένα άλλο θέμα. Από φέτος θα υπάρξουν περιφερειακές μεταρρυθμίσεις στην Τσεχία, στη Λουδανία, στην Λετονία. Θα υπάρχουν δύο περιφέρειες και οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών περιφερειών είναι πάρα πολύ σημαντικές. 100% στήριξη από την μία σε μία από αυτές τις περιφέρειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πολύ λιγότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ θα υποβάλω την πρότασή μου. Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο και σωστό να υπάρχουν περικοπές σε κράτη-μέλη που έχουν φτάσει στο μέσο όρο του 75%. Τα κράτη-μέλη που έχουν φτάσει στο 75%, οι περικοπές πάνω από 20% είναι υπερβολικές. 10% όχι παραπάνω. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου αφορά την χρηματοδότηση, το επίπεδο της χρηματοδότησης που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 15% για άλλες είναι 45% εάν ένα κράτος μέλος, παραδείγματος χάρη, έχει διαφορετική κατανομή στις περιφέρειές τους, θα θέλαμε να υπάρχει περισσότερη σύγκληση και περισσότερες δυνατότητες να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αυτές τις διακυμάνσεις και τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών. Και από ό,τι διαβάζω εδώ στο έγγραφο αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και τους αριθμούς. Λαμπρά, σας ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Μπούντα που είναι ο σκιώδης Τα δικά του σχόλια μεταφέρω γιατί εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη με τις λεπτομέρειες. Η πρόταση στόχο έχει να μειώσει το διοικητικό άκθος για τους δικαιούχους και τους ε, φορείς διαχείρισης, κρατώντας ένα υψηλό βαθμό νομιμότητας και ε, κανονικότητας με ένα κανονισμό περί κοινών διατάξεων για 7 ταμεία. Όμως, όπως επισήμανε η συγγήτρια, αποκλείεται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης ε, της Υπέθρου. Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε την αρχή επικουρικότητα για την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των γεωργών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει προσθέσει ε, διοικητική περιπλοκότητα σε επίπεδο παραγωγού. Η Επιτροπή μας ε, ε, έχουμε, έχει ήδη επισημάνει στην έκθεση Dorfman για το μέλλον της Γεωργίας ότι δεν θα πρέπει η επικουρικότητα να αυξάνει την ε, γραφειοκρατική περιπλοκότητα της κάπου Οποιαδήποτε επιπλέον επικουρικότητα θα πρέπει να στηρίζεται από ένα ε, ισχυρό κοινό κανονιστικό πλαίσιο. Είμαστε υπέρ της πρότασης ηγητρίας να, να παραμείνει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ανάπτυξης ε, της υπαίθρου στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, τοπικές ε, αναπτυξιακές στρατηγικές γιατί αυτές είναι που έχουν δώσει αυτά αποτελέσματα και επίσης οι κοινότητες ενδιαφέρονται για τοπικές δράσεις θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη δική τους εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα στη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαγκίνες, η κυρία Αγγιλέρα και μετά κύριος Δαντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω για την γνωμοδότηση της κυρία Ζωανά ότι συμφωνώ με το πιο σημαντικό που είναι η γνωμοδότηση Επιτροπής Γεωργίας θα πρέπει να αφορά τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών ταμείων και κυρίως ε, από δύο σκοπιές που πολύ σωστά τις επισημαίνει η, η Φυσικά διαφωνούμε με την δημοσιονομική περικοπή και κυρίως ε, συμφωνούμε με την ε, καταγγελία των μεγάλων περικοπών στον, στο Περιφερειακό Ταμείο Επίσης, η ΚΑΠ εξεκολουθεί να έχει τους ίδιους πόρους με το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και θέλουμε να τους διαφυλάξουμε που δεν θα δεχτούμε μείωση και θα δώσουμε μάχη όχι μόνο στη συζήτηση για την ΚΑΠ αλλά και στη συζήτηση για τα διαρθρωτικά ταμεία για να αποφευθούν πε, περικοπές. Επίσης, στον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, γιατί αποκλείστηκε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη. Ε, δεν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Θα προτιμούσα το Γεωργικό Ταμείο μαζί με τα υπόλοιπα ταμεία που επίση θεωρούνται διαρθρωτικά. Γιατί πρόκειται για ταμεία που προσπαθούν να εξαλείψουν τι ανισότητες μεταξύ ζωνών και περιφερειών και εδαφών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η είμαστε υπέρ του μεγαλύτερου συντονισμού και εναρμόνιση. Γι' αυτό θέλουμε και το Γερικό Ταμείο να μπει στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Αυτός, αυτή η αφαίρεση του Γερικού Ταμείου από τον κανονισμό και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι άστοχη κατά τη γνώμη μου. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες. Έχουμε και ένα άλλο στοιχείο. Τα διαρθρωτικά ταμεία χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων ε, για τη διαφορά της συγχρηματοδότησης. Ε, αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Ροπέλα αντίθετε συγγνώμη, Θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά επίπεδα συγχρηματοδότηση στο μέτρο που έχουμε διαφορετικά κατακεφαλήν εισοδήματα στα κράτη-μέλη. Στο μέτρο που δεν έχουμε μια ισότητα στο κατακεφαλήν εισόδημα και στην ποιότητα ζωή σε όλε τι ευρωπαϊκέ περιφέρειε, δεν θα πρέπει να έχουμε σύγκληση ούτε στο ποστό χρηματοδότηση και στι διαρθρωτικέ ενισχύσει. γιατί ε, δεν μιλούμε εδώ για τις άμεσες ενισχύσεις του Γεωργικού Ταμείου, αλλά το Γεωργικό Ταμείο και τα Διευθυντικά Ταμεία στόχο έχουν να βγάλουν από, το περιθώριο, να καταπολεμήσουν την περιθωριοποίηση στα ευρωπαϊκά εδάφη και περιοχές. Γι' αυτό καλύτερα να είναι το Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης Υπαίθρου εντός του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και να μην αποκλείεται. Συμφωνώ με τις τροπολογίες της ε, κυρία Ζωανά που ξαναβάζει το Γεωργικό Ταμείο στον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, που ούτως ή άλλως δεν είχε νόημα να αποκλειστεί από την αρχή. Ο κύριος Δαντά. Ευχαριστώ. εξ ονόματος ε, του συναδέλφου Μίλλερ. Σας και του οριζόντιου αυτού κανονισμού, παίρνω το λόγο. Διαφωνώ. Παρόλο που κατανοώ αυτά που ακούστηκαν. Πρέπει να βρούμε μια μέση λύση, πιστεύω. Αν είμαστε καθαρά, αν θέλετε, υπό την οπτική των περιφερειών και της δημόσιας ε, άσκησης πολιτικής, Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη χρηματοδότηση, αλλά τελικά ποιος υποφελείται από το ταμείο, από το ΠΕΝΤΕΡ. Και αν το διατηρήσουμε στον κανονισμό με τα άλλα ταμεία, γίνεται πιο περίπλοκο διοικητικά το σύστημα, διότι υπάρχει πρώτος πυλώνας με μία λογική και ο δεύτερος πυλώνας με μία διαφορετική λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς εδώ στην Επιτροπή μας προσπαθούμε να διευρύνουμε την απλοποίηση να εναρμονίσουμε. Δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε 100%. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά δεν γίνεται 100%. Θα πρέπει όμως να στηρίξουμε τα συμφέροντα των αγροτών. Υποβάλλουν ένα φάκελο για χρηματοδότηση και αυτός ο φάκελος ελέγχεται. Το γεγονός ότι το ΦΕΝΤΕΡ έχει τελείως διαφορετικούς κανόνες από αυτούς του πρώτου πυλώνα περιπλέκει σημαντικά τα πράγματα για αυτούς που υποβάλλουν αιτήσει χρηματοδότησης, δηλαδή για τους γεωργούς. Βεβαίω υπάρχει μια κατανομή μεταξύ Φέντερ, Φέαντερ κτλ. Αλλά προ συμφέρον, επαναλαμβάνω, των γεωργών, σε αυτόν τον οριζόντιο κανονισμό θα πρέπει να οδηγηθούμε προς μια ομοιογενοποίηση όλων αυτών των κανόνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μισελ. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ τα δική μου απόψη. Δεν έχω ενημερωθεί απόλυτα για αυτό το φάκελο, αλλά έχω και εγώ κάποια θέματα που με απασχολούν βάσει όσων είπε ο Μισελ. Αλλά κύριε Ντόρφμα, ζητήστε το λόγο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις. Πριν από ένα χρόνο συζητήσαμε για τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις της και το θέμα είναι πόσο ενσωματώνεται και πόσο λαμβάνουμε υπόψη μα τα θέματα που αφορούν την περιφερειακή πολιτική. Εδώ στην Επιτροπή Άγκρη ήμασταν πάντα πολύ αυστηροί όσον αφορά το οπτικό πεδίο το, στο οποίο εμείς στοχεύουμε. Γεωργική πολιτική και κατά πόσο αυτή η γεωργική πολιτική ενσωματώνει στοιχεία της περιφερειακής πολιτικής που στοχεύουμε. Εγώ παραδείγματο χάρη και στη δική μου περιοχή έχω πάρα πολλές περιπτώσεις όπου βεβαίως κάποια χρηματοδότηση έμεσα φτάνει στους γεωργούς από τα ταμεία περιφερειακής πολιτικής και επηρεάζει φυσικά την περιφερειακή πολιτική. Το θέμα είναι ότι άλλη είναι η περιφερειακή πολιτική και θα πρέπει να μην ξεχνάμε τη βασική μας κατευθυντήρια γραμμή και να μην ξεπερνάμε την ημερήσια διάταξη. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να υπερασπιστούμε ε, ο δεύτερος πυλώνας να παραμείνει καθαρά θέμα της αγροτικής πολιτικής. Αν ναι, τότε και εδώ θα πρέπει η εισηγήτρια να ξαναδεί την γραμμή της και όλες τις τροπολογίες. Θα πρέπει να υποβάλουμε νέες τροπολογίες. Θα πρέπει να ξαναδούμε δηλαδή και να ξανασυζητήσουμε το θέμα του δεύτερου πυλώνα και του μέλλοντος της εξέλιξης του δεύτερου πυλώνα. Γιατί πραγματικά σκοπός μας δεν είναι εδώ να περιοριστούν τα κονδύλια που φτάνουν στους αγρότες. Ευχαριστούμε, Χέρμπερτ. Πριν δώσω το λόγο και πάλι ε, στη συνάδελφα Ζωάννα, να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Εδώ βρίσκεται η Διευθύντρια κυρία Ρομάνσκα. Παρακαλώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Λέγομαι Ρομάνσκα από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγια. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής ε, και με το νέο πλαίσιο που προτείνουμε. Κατά την προετοιμασία της αμαθητικής πρότασης για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προκύπτουν από το Brexit. Και αυτό χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες δύσκολες επιλογές. Η πολιτική συνοχή έχει περικοπεί περισσότερο από την κυνηγιορική πολιτική. Και γι' αυτό έπρεπε να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε συνοχή, συνέπεια και σαφήνεια και για τις δημόσιες αρχές αλλά και για τους δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της συγγετρίας, της συντάκτης γνωμοδότησης. Ένας από τους βασικούς κλάδους των, της συνέργειας είναι στην κοινότητα, τη, το, τοπικές κοινότητες για την ανάπτυξη. Και αυτό διαφυλάσσεται και για το 2020. Σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και την προβλεψιμότητα υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις, Συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους από την Κοινική Διάθεση Γεωργίας, ώστε να εξασφαλίσουμε συνέπεια και ενάρια μεταξύ του, κοινού, του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και του κανονισμού περί κοινή γεωργικής πολιτικής, γιατί θέλουμε να έχουμε αρμονική εφαρμογή των κανόνων επιτόπου. Και επειδή αναμένεται η μεγάλη γενική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αν αναγκάζουμε τους, ε, τις δημόσιες αρχές και τους δικαιούχους να με, μεταπηδούν από τον ένα κανονισμό στον άλλο συχνά, θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση, κάτι που θα παρεμποδίσει και την εύρυθμη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Και επανέρχομαι στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, CPR. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ροπέ, όντως οι περικοπές είναι σημαντικές, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι παρόλο που κάποιες χώρες μέλη έχουν χάσει περίπου 23% των κονδυλίων τους, στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, 2014-2020, κάποιες χώρες είχαν χάσει μέχρι και 45% των κονδυλίων. Οπότε η απώλεια στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μικρότερη. Και γι' αυτό κρίνουμε την πρότασή μας ισορροπημένη. Μάλιστα, λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι κάποιε χώρε ε, σημείωσαν εντυπωσιακή πρόοδο στην κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τώρα το νέο διαχωρισμό των περιφερειών στη Λιθουανία, Ουγγαρία Πολωνία, η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζεται στα πιο ενημερωμένα στοιχεία ε, μέχρι το 2016 και γι' αυτό ε, ο νέος χαρακτηρισμός των περιφερειών και ο νέος διαχωρισμός δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη μέχρι τώρα. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο συγχρηματοδότηση, όντω μειώθηκε το ποσοστό συγχρηματοδότηση. Αρχικά είχε αυξηθεί λόγω κρίση και τώρα που βρίσκεται και πάλι σε πορεία ανάπτυξη η ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία, ζητούμε από του εθνικού και τοπικού προπολογισμού ε, να αναλάβουν τι ευθύνε του και να αυξήσουν την συμμετοχή τους ε, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά και αν έχετε και άλλες απορίες είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τον τελικό λόγο στη Μαρία Γκαμπρέλα Τζοάνα. Όχι. Οκ. Ε, μπορείτε να ε, κλείσετε τη συζήτηση, Τζοάννα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Και όπως είπα, 26 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Περιμένω με ανυπομονησία τις τροπολογίες σας και θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινήσεις. Δεν πρόκειται για την εφαρμογή, διαφοροποιημένη εφαρμογή μεταξύ των δύο πυλώνων. Αυτό που θα γίνει είναι η εφαρμογή των κανόνων της κοινή αγροτικής πολιτικής και θα απαντήσω στο συνάδελφο ότι όλοι οι κανόνες του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις ήδη εφαρμόζονται για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν ξέρω αν δεν έγινε κατανοητό το κείμενό μου. Επαναλαμβάνω, περιμένω τις τροπολογίες σας για να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταξύ αναφέραμε την ημερομηνία για τις τροπολογίες. Κλείνουμε το 5 και πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο σημείο 6. Αφορά και πάλι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Η συγητής είναι ο Τζέιμς Νίκολσον και του δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ, Τζέιμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εγκρίνουμε αυτή την ε, έκθεση. Ε, ε, εδώ οι αποφάσεις αυτές θα, θα αφορούν τους γεωργούς μας και τις αγροτικές κοινότητες όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Θα μείνω συνοπτικός. Θέλουμε η περιφερειακή ανάπτυξη να έχει την ίδια προσοχή με την αστική ανάπτυξη. Πολλοί γεωργοί ε, χρειάζονται, εργάζονται και online τώρα και χρειάζονται πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες που υπογραμμίζουν ε, τη σημασία των κοινών δραστηριοτήτων και θέλω ε, να ε, τονίσω το θέμα των επενδύσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Επίσης έχω υποβάλλει τροπολογίε ε, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στι γεωργικές περιοχέ, στις αγροτικές περιοχές, την εκπαίδευση, την κατάρτιση για διάφορε δεξιότητε να μην είμαστε εστιασμένοι μόνο στι αστικέ περιοχέ. Οι αστικέ περιοχέ θεωρείται ότι δίνουν ε, δουλειέ, αλλά μην ξεχνάμε και τι γεωργικέ ε, αγροτικέ περιοχέ που έχουν πιστεύω ίδια σημασία και σπουδαιότητα όπω και οι αστικέ περιοχέ σε θέματα δημιουργία θέσεων εργασία. Οπότε πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό για την καινοτομία και τις καινοτόμες ε, ε τεχνολογίες στο 65% από το 60%. Πιστεύω είναι μικρή αυξησία αλλά θα δείξει ότι υποστηρίζουμε τις γεωργικές τεχνολογίες. Αναμένω να συνεργαστώ με τους κοιόδης και όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι πολύ στενά τα περιθώρια για την υποβολή των τροπολογιών, αλλά αυτό έχει γίνει ώστε να, γίνει, δοθεί η γνωμοδότησή μας πριν ε, έγκαιρα στην Επιτροπή ε, Ρέτζι. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό, πιστεύουμε, και θα γίνει όλο και πιο σημαντικό καθώς θα αρχίσουμε να συζητάμε τα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Ροπέ, πάλι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αδικαιολόγητη μείωση της χρηματοδότησης είναι απαράδεκτη. Δεν φταίνουν ε, το Ταμείο Συνοχής ή το Περιφερειακό Ταμείο για το Brexit. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δείξουν αλληλεγγύη και να Ανεβάσω τη συμμετοχή του στο 1,36% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο για να αντιμετωπίσουμε τι νέε προκλήσει. Χωρί όμω να ξεχνούμε και τι παλιέ προκλήσει. Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στι νέε προκλήσει και να αμελούμε τι παλιέ. Είναι άδικο αυτό. Θα πρέπει να το διορθώσουμε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Νίκολσον ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθεί περισσότερο για τις περιφέρειες. Ε, χρειαζόμαστε κάποια περιφερειακά κέντρα που διαχειρίζονται τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου και που έχουν πολύ μεγαλύτερη ε, πρωτοβουλία, δείχνουν πολύ μεγαλύτερη πρωτοβουλία και δεν θα πρέπει να απορροφώνται περισσότερα κονδύλια στα αστικά κέντρα, στις αστικές περιοχές. Θα πρέπει να προβλέψουμε ένα ποσοστό το κονδυλίου που θα πηγαίνουν σε αγροτικές περιοχές. Γιατί ε, τα περιφερειακά κέντρα, τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκταμιεύουν το 90% των κονδύλιων, ενώ οι μικρές πόλεις, ή αγροτικές ζώνες μένουν με τα ψίχουλα. Και τους λένε υποβάλλετε τα έτοιμά σας στο πρόγραμμα Leader. Τι γίνεται με το πρόγραμμα Leader λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μόνο 5% για το Leader από το Περιφερειακό Ταμείο. Θα προτιμούσαμε 10%, όχι μόνο 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μόνο το 5%, που είναι 40% σε σχέση με αυτό που είχαμε το 2020. Έγινε μείωση κατά 2,5% υποδιπλασιασμός μάλλον των κονδύλων αυτών, δυσκολία πρόσβασης από τις αγροτικές ζώνες στα κονδύλια, οπότε το πλήγμα για τις αγροτικές ζώνες είναι ακόμη μεγαλύτερο. Και μετά διαρριγνύουμε τα ημάτια μας γιατί δεν έχουμε νέους γεωργούς, γιατί δεν πηγαίνει νεολαία στην Ήπεθρο για να ζήσει. Μα πώς θα προσελκύσουμε νέους στην Ήπεθρο και στη Γεωργία αν δεν τους υποστηρίξουμε. Το πρόγραμμα Leader ε, λειτουργεί εύρυθμα σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν είχαμε ποτέ μομφές εναντίον του. Το πρόγραμμα Leader έχει απτά και θετικά αποτελέσματα για τους συμπολίτε μας και μάλιστα ενεργοποιούνται σε αυτό και οι τοπικές αρχές, τοπικές ομάδες και συνεταιρισμοί, το, τοπικές επιχειρήσεις και εξασφαλίζεται και καλύτερος έλεγχος με μεγαλύτερο περιορισμό του ποσοστού σφάλματος. Στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο χρειαζόμαστε ένα είδος προγράμματος LEADER. Θέλουμε παρόμοιο πρόγραμμα να χρησιμοποιείται και στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο, σαν το LEADER, το επιχειρήσεις, ε, κοινότητες, τοπικές αρχές να μπορούν να συμμετέχουν στο Ταμείο και να μπορούν να χρηματοδοτούν τις ιδιαίτερες τους ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Στίορ Ντάκνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντας τα όσα είπε ο κύριος Ρόπε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του. Τα ταμεία αυτά φαίνονται πολύ δύσκολα ε, όσον αφορά την πρόσβαση των αγροτών σε αυτά. Εκτός από το Ταμείο Leader, ακούμε γι' αυτό περισσότερο από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ότι έχουν πρόσβαση. Ω ιδέα, η ύπαρξη αυτών των ταμείων ακούγεται καταπληκτική. Αλλά και, και ελπίζω, Τζιμ, να επανέλθει σε αυτά που λέω και εγώ, γιατί κάνει τη δουλειά αυτή εδώ και καιρό και εκπροσωπεί και τη Βόρεια Τζιμ, Αυτά τα ταμεία περιφερειακή ανάπτυξη και το Ταμείο Συνοχή θεωρεί ε, ότι έχουν εύκολη πρόσβαση όσον αφορά του αγρότε στη δική σου εκλογική περιφέρεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Στιουάρτα. Τώρα να δώσω ξανά το λόγο στην Επιτροπή. Στην Δόκτωρ Ρομάνσκα. Παρακαλώ. Thank you ε, Καταρχήν, στηρίζει το Ταμείο τη Επαρχία και φυσικά δεν υπάρχουν, την δεν υπάρχουν νέοι περιορισμοί. Εμείς αποφασίσαμε να στηρίξουμε την τοπική ανάπτυξη με πολύ συγκεκριμένους στόχους ε, για αυτήν, πέντε, χάρη στο Περιφερειακό Ταμείο και στο ΕΚΤΑ θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες ε, περισσότερο και πιο αποτελεσματικά. Η Επιτροπή έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις ε, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία της ε, στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θελήσαμε να στηρίξουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και πολύ φοβάμαι ότι αν θελήσουμε να καλύψουμε περισσότερες δραστηριότητες, δεν θα στοχεύσουμε σωστά όπως θέλαμε. Γι' αυτό και ακριβώς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε επικαλύψεις μεταξύ της στήριξης των διαφορών ταμείων, παραδείγματος χάριν, το άρθρο 6 του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, όπως είπε και ο εισηγητής, στοχεύει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε περαιτέρω σύγχυση και ε, για αυτούς που θέλουμε να υποφεληθούν από αυτή την στήριξη, αλλά και από τις διοικητικές αρχές. όσον αφορά το θέμα της ε, ευρυζωνίας. Και εδώ θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και πιστεύουμε ότι σε κάποιες περιοχές όπου είναι πολύ αργή, πολύ αργά τα δίκτυα, όπου είναι πολύ δαπανηρά, θα πρέπει να επενδυθούν περισσότερα κονδύλια. Σήμερα Ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο με τους παρόντες κανονισμού να αυξηθεί η χρηματοδότηση όσον αφορά παρέμβαση δημόσιων ασχολών. Αυτές είναι οι περιοριστικές διατάξεις που υπάρχουν ακόμα στα θέματα ευρυζώνειας. Τζιμ, τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θέμη και εγώ σύντομος. Υπάρχει κάποια σύγχυση μεταξύ του Ταμείου Συνοχή και του Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. Και ποιοι είναι οι σκοποί των δύο ταμείων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύγχυση. Το πρόγραμμα Leader, κατά την άποψή μου, υπήρξε ένα από τα καλύτερα προγράμματα που ποτέ ψήφισαν οι Βρυξέλλε. Χρησιμοποιήθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικά από πολλές ε, γεωργικές κοινότητες, πολλούς ε, πολλέ οργανώσει αγροτών, συνεταιρισμού και χρησιμοποιήθηκε σε εποχέ στη Βορεια Ιρλανδία για μεγάλο κομμάτι τη διασυνοριακή συνεργασία. Ε, στα σύνορα Βορρέ και Ιρλανδία και Δημοκρατία τη Ιρλανδία έφερε ανθρώπου κοντά οι οποίοι ουδέποτε θα είχαν έρθει χωρί αυτό σε επαφή. Είμαι μεγάλο υποστηρικτή λοιπόν του προγράμματο Leader και μπορούμε να το αναπτύξουμε και να το εξέλιξουμε παραπάνω. Δεν θέλω να χαθεί το Leader. Αλλά οι αγρότες ε, που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Ξέρετε, κοιτάξτε, όλα τα προγράμματα, ανεξαρτήτως του ποιο είναι το πρόγραμμα, όσοι προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση αυτά σας λένε πάντα το ίδιο, είναι δύσκολη η πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι είτε μιλάμε για διαχείριση σε τοπικό επίπεδο είτε για διαχείριση από τις Βρυξέλλες, κανένας δεν μπορεί απλά να δώσει λευκή επιταγή σε οποιονδήποτε ε, και να αρχίσει να μοιράζει λεφτά χωρίς κάποιο έλεγχο έστω και ελάχιστο. Και αυτό που έχω να πω στον κύριο Αγνιού, ναι, πράγματι δυσκολεύονται και σίγουρα ε, από εκεί που έρχομαι εγώ στη Βόρεια Ιρλανδία οι Γεωργοί ίσως να μην τα πάνε τόσο καλά όσο στην Ανατολική Αγγλία που αυτός ε, προέρχεται αλλά χρειάστηκε να το κάνουμε αυτό, να υπάρξει κάποια πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια με κάποιο τρόπο. Ίσως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία, ε, η κύρια ίσως ε, να μην είχε τόσο αρκετή πρόσβαση και να θύμωσε γι' αυτό και να έχουμε γι' αυτό το Brexit, αλλά εμείς είχαμε πρόσβαση, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος σε κάποιο βαθμό. Εγώ γνωρίζω του συναδέλφου μου, του ε, Γιώργου πολύ καλά και θα ήθελα να είναι τα πράγματα όσο το δυνατόν ευκολότερα. Αλλά ξέρετε, του ξέρω ε, επίση καλά και ξέρω ότι όπου υπάρχουν λεφτά θα πάει άλλο να τα πάρει. Ξέρετε, η πρόσβαση των αγροτών ε, τελικά στα χρήματα αυτά οδηγεί στην καλή του χρήση και υπάρχουν ωφέλη ορατά. Και αλλά είμαι έτοιμο να ακούσω τα όσα θέλετε να πείτε και άκουσα και τα όσα είπε και ο κ. Ρόπα και όσα που όλοι οι υπόλοιποι στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Ε, ευχαριστώ να ακούσω όλε τι απόψει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστούμε, Τζιμ. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου. Θα θεωρήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. Να σα υπενθυμίσω, είναι πολύ σημαντικό. 1η Οκτωβρίου να βρισκόμαστε όλοι στην, συνεδρίαση, στην έκτακτη συνεδρίαση τη Επιτροπή, όπου θα ψηφίσουμε την οδηγία μας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και εύχομαι ειλικρινά να επιτύχουμε ευρεία πλειοψηφία από όλες ομάδες. Ευχαριστώ σε όλους, καλή δουλειά και θα τα πούμε στο Στρασβούργο.